Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, να ξεκινήσουμε. Έχετε δει την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, εγκρίθηκε. Δύο ανακοινώσεις του Προέδρου. Σας υπενθυμίζω ότι όλες οι γλώσσες που χρειάζονται τα μέλη της Επιτροπής μας είναι διαθέσιμες. Έχετε λάβει τα αναγκαία έγγραφα. Υπενθυμίζω, όπως ξέρουν οι προσκεκλημένοι μας, ότι η συνεδρίασή μας αυτή είναι δημόσια, όπως όλες μας οι συνεδριάσεις, οπότε υπάρχουν θέσεις για το κοινό και οι συζητήσεις μας μεταδίδονται ζωντανά μέσω web streaming στο ίντερνετ. 3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασής μας της 1ης Ιουνίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι ενεκρίθησαν και μπορούμε να περάσουμε απευθείας στο σημείο 4, ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους ορισμένων ε, εταιριών, τριών συγκεκριμένα πολυεθνικών, οι δύο είναι πιο πολυεθνικές από την τρίτη, για το θέμα μας. Πριν τους δώσω το λόγο, υπενθυμίζω το πλαίσιο στο οποίο θα διεξαχθεί η ακρόαση σήμερα το πρωί. Η Επιτροπή μας είναι προσωρινή Επιτροπή για να διερευνήσει τις πρακτικές των φορολογικών αποφάσεων και άλλων νομοθετημάτων ή πρακτικών που μπορούν να διασφαλίζουν προνομιακή μεταχείριση και να θίγουν τον θεμητό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και παγκόσμια. Η Επιτροπή μας προσπαθεί να συλλέξει τις μέγιστες δυνατές πληροφορίες για αυτές τις πρακτικές και να κάνει πολιτικές συστάσεις παράλληλα με τις εργασίες που γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα για το θέμα αυτό από τον ΟΟΣΑ, υπό την ηγεσία του ΟΟΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα δράση που ο Πρόεδρο Γιούγκερ θα μα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα. Θα έρθει εδώ να μα τις παρουσιάσει. Να μα το παρουσιάσει το πρόγραμμα δράση. Στα πλαίσια τη συλλογή πληροφοριών έχουμε στείλει αποστολέ Ενημέρωση ε, στις έξι χώρες που θεωρούσαμε ότι είναι οι πιο προβληματικές, πέντε εντός της Ένωσης και στην Ελβετία. Έχουμε ακούσει πολλές προσωπικότητες που έχουν αρμοδιότητα για το θέμα αυτό είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στον ΩΣΑ είτε είναι εμπλεκόμενοι φορείς κατά τον α τρόπο. Για παράδειγμα, ε, μία ένωση δημοσιογράφων που είναι αρμόδιοι για τα LuxLeaks και τα Leaks. Επίσης αυτοί οι οποίοι έχουν καταγγείλει ορισμένες τέτοιες πρακτικές και ορισμένες εταιρείες λογιστικού ελέγχου και συμβουλών που ε, δίνουν συμβουλές ε, στους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις για την φορολογική του στρατηγική. Λεγόμενοι μεγάλοι τέσσερις. Τέσσερις μεγάλοι. Οι αρμόδιοι των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου θέλησαν να ακούσουν και τι έχουν να μας πούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι πολυεθνικές. Και ευχαριστώ τους εκπροσώπους των τριών επιχειρήσεων που είναι παρούσες σήμερα. Θα υπάρξουν και περαιτέρω συζητήσει, αυτή είναι η πρώτη πρέπει ε, να διαπιστώσω ότι κάποιες χώρες ε, ε, από πλευράς φορολογίας βοηθάνε και άλλες δεν βοηθάνε. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς επιχειρήσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις δείχνουν καλή διάθεση να συνεργαστούν, ενώ άλλες όχι. Σήμερα βέβαια αυτές που είναι παρούσες δείχνουν θετική διάθεση. Θα πρέπει να αποφασίσουμε, αλλά όχι σήμερα, ποιε θα μπορούσαν να ήσαν οι επιπτώσει για τι σχέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τι επιχειρήσει που δεν δείχνουν διάθεση συνεργασία. Αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Αλλά ήθελα να το αναφέρω. Σήμερα λοιπόν έχουμε εδώ την κυρία Ναταλή Μόνιετη που είναι επικεφαλής ε, της ε, φορολογικής υπηρεσίας της Total η Total νομίζω είναι η μεγαλύτερη γαλλική εταιρεία από πλευρά κύκλου εργασιών και η τέταρτη επιχείρηση από πλευρά κύκλου εργασιών ε, στον τομέα των ίδρογων ανθράκων παγκόσμια που έχει δραστηριότητες ε, σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου τουλάχιστον ε, σε όσες μπορεί κανείς να εξαγάγει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο κύριος Μάρτιν Μακιούν επίσης είναι επικεφαλής της υπηρεσίας της φορολογικής υπηρεσίας SSE που έχει μια σειρά από επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας και δραστηριότητες ιδιαίτερα στη Σκωτία. Και έχουμε επίσης τον κύριο Κριστιαν Κομολετιγμό που είναι υπεύθυνο για τα φορολογικά στην BNP Paribas, τον όμιλο BNP Paribas. Ε, μία από τις μεγαλύτερες γαλλικές και ευρωπαϊκές τράπεζες που έχει δραστηριότητες σε 75 χώρες. Οι τρεις αυτές επιχειρήσεις έχουν ένα κοινό στοιχείο. Πρώτον, δέχτηκαν να συνεργαστούν μαζί μας. Δεύτερον, δεύτερον, ένα από τα σημαντικά πολιτικά θέματα που θέλουμε να εξετάσουμε και που το συζητάμε και θέλουμε να κάνουμε προτάσεις γι' αυτό και στον ΩΣΑ είναι οι εκθέσεις αναχώρα. εφαρμόζεται στους τομείς ε, δραστηριότητάς τους. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η άποψή τους για το σύστημα αυτό. Στρέφομαι προς ε, τους εισηγητές μας. Προβλέπουμε να κάνουν εισαγωγές ε, πρώτα απ' όλα οι εμπειρογνώμονές μας. Θέλουν τίποτα να πούν οι εισηγητές μας. Ούτε η Λίζα ούτε ο Μικαέλ βλέπω. Ωραία, θα μας κάνουν μια εισαγωγή με τη σειρά που τους ανέφερα. Σας παρακαλώ να μην ξεπεράσετε ο καθένας 10 λεπτά για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μία ανταλλαγή έρωτα αποκρίσεων. Θα είμαι αμήλικτος. Στο λεπτό θα κόβω το λόγο. Και η κυρία Μονιετή θα μιλήσει πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην, που δώσατε στην, στον Όμιλο Total να έρθει εδώ στην Επιτροπή σας να μιλήσει. Να σας παρουσιάσω ποιος είμαι. Είμαι η Διευθύντρια για τα φορολογικά θέματα εδώ και δύο χρόνια της Total. Πριν από αυτό ήμουνα ε, υπεύθυνη για τη διεθνή φορολογία, ε, το το σύνολο της καριέρας μου το έχω αφιερώσει στην Total 17 χρόνια για τα θέματα τα φορολογικά κυρίως. Να σας μιλήσω λιγάκι για τον όμιλο Total και για την πολιτική του για τα φορολογικά. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί νομίζω ότι έχετε λάβει την παρουσίασή μας. Όπως είπε και ο πρόεδρος Λαμασούρ, η Total είναι η τέταρτη ε, εταιρεία πετρελοειδών παγκοσμίω ε, στο χρηματιστήριο. Είναι η πρώτη εταιρεία που είναι στο χρηματιστήριο το 2014 ε, η Total είναι η ΕΣΑ, ε, είναι η βασική εταιρεία του ομίλου, δημιουργήθηκε στο, το 2024. Ε, έχουμε 903 θηγατρικές, 130 χώρες και τον κατάλογο με το ποσοστό των μετοχών καθώς και τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα τους ε, υπάρχει στα βασικά μας έγγραφα και στην ιστοσελίδα μας. Πολύ σύντομα, η Total είναι μια εταιρεία πετρολιδών ε, που έχει ε, δραστηριότητες όλων των, τους τομείς και στις ανάντι δραστηριότητες, δηλαδή αναζήτηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, αλλά και στις κατάν δραστηριότητες, δηλαδή στις παραδοσιακές δραστηριότητες, δίληση, πετροχημία, ε, ειδική χημεία, ε, διανομή ε, των προϊόντων και διεθνές εμπόριο του αργού πετρελαίου και του πετρελαίου. Η Total είναι σημαντικός παράγοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είμαστε το νούμερο, 2 παγκόσμια της αεολικής ενέργειας με τη SunPower, την Αμερικάνικη εταιρεία που κατέχουμε το 60% αυτής. Επίσης η ομάδα μας έχει επίσης 100.000 συνεργάτες 100 και τους 33 στη Γαλλία. Κάποια βασικά στοιχεία. Το 2014 η Total υλοποίησε 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια ε, καθαρού αποτελέσματος ε, ε και ο τζίρος ήταν 236 εκατομμύρια δολάρια. Η Total την ίδια χρονιά ε, φορολογήθηκε στα κέρδη της 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι το 53% ε, ο φορολογικό τελεστή. Ε, Επίση, θα πρέπει να προσθέσουμε 5 δισεκατομμύρια δολάρια άλλων φόρων ε, ειδικών για το πετρέλαιο ε, και την παραγωγή του πετρελαίου. Οι διάφοροι τομεί δραστηριότητα και το ειδικό του βάρο. Ο ανάντι τομέας έχει τις δραστηριότητες της αναζήτησης ε, και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και είναι ο πιο βασικός τομέας μας ε, κεφαλαϊκά και, ε, και των αποτελεσμάτων, γιατί είναι περίπου το 80% της αξίας των, των στοιχείων του ενεργητικού και των 26,5 δισεκατομμυρίων επενδύσεων που κάναμε το 2014. Είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι μακροπρόθεσμη, και φορολογικά είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσω. Η χημική δίληση έχει τις δραστηριότητες ε, της πετροχημίας, ε, δίλησης και εξειδικευμένης χημίας και είναι κάτι παραπάνω το 10% των ε, κεφαλαίων που μας απορροφά. Η Total έχει συμμετοχή σε 21 δηληστήρια. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι ο πρώτος δηληστής στη Δυτική Ευρώπη. Ε, το marketing και οι υπηρεσίες έχει όλες τις δραστηριότητες εμπορίας, ε, ε, πετρολοειδών, νέων ενεργειών που υπάρχουν πολύ έντονα στην Ευρώπη και που είναι Επίσης, ε, ο πρώτος διανομέας ε, ε, πετρελοειδών στην Αφρικανική Ήπειρο και είναι 15.000 βενζινάδικα το 2014, το τέλος του 2014. Αυτή είναι μια γρήγορη παρουσίαση της Total για να μπορέσετε να καταλάβετε λιγάκι τον διεθνή χαρακτήρα της εταιρείας και το μέγεθος του ομίλου. Σε ό,τι αφορά την φορολογική του κατάσταση, η Total είναι η γαλλική εταιρεία που πληρώνει τις περισσότερες, τους περισσότερους φόρους επί των κερδών Έχουμε διαφθορτικό φορολογικό συντελεστή πάνω από 50%, 53% το 2014, 58% μερικές χρονιές και επομένως το 2014 ε, ε, πληρώσαμε πάνω από 8 δις δολάρια. Να τονίσω ότι είμαστε μια βιομηχανική ε, εταιρεία, ένας βιομηχανικός όμιλος, όπως παρουσίασα στην αρχή. Είμαστε Ανήκουμε στη βαριά βιομηχανία φυσικά. Δεν ε, είμαστε στις άλλες, ε, στις υπηρεσίες ε, ή σε οτιδήποτε άλλο. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία είναι σημαντικό γιατί τα κέρδη μας συνδέονται άμεσα με το υπέδαφος, με το έδαφος όπου βρίσκονται τα αποθέματα, οι πλατφόρμες μας, τα εργοστάσια μας και δεν μετεγκαθίστανται λοιπόν. Λόγω αυτού ο όμιλός μας πληρώνει τις, τους φόρους ε, επί των κερδών εκεί όπου υλοποιούνται τα κέρδη, δηλαδή όπου παράγονται ε, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπου οι φορολογικοί συντελεστές είναι πολύ ψηλοί, πάνω από τους συνήθεις φορολογικού συντελεστές, ε, παραδείγματο χάρη 78% στην Ορβηγία, 76,5% στην Κάμπια, 85% επί του εδάφου της Νιγήριας, 50% υπεράκτεια στην Αγγόλα έχουμε δηλαδή πολύ πιο υψηλού φορολογικούς συντελεστέ από ό,τι συνήθως. Πολύ λογικά λοιπόν το 2014 η Αφρική ήταν 55% ε, του φόρου μας, ε, ε, η Ευρώπη 24%, κυρίως στην Νορβηγία και το, τους υπόλοιπους φόρους τους πληρώσαμε στον υπόλοιπο κόσμο 20%. το διεθνές μας εμπόριο του αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου αφορά ε, προϊόντα τα οποία έχουν μπει σε διεθνείς αγορές, ε, διεθνή χρηματιστήρια. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να καθορίσουμε όπως να είναι τις τιμές μεταβίβασης. Και το περισσότερο πετρέλαιο που παράγουμε πουλιέται διεθνώς ας πούμε και αγοράζεται από τρίτους πάλι σε διεθνείς αγορές. Ε, πάντα σε τιμές χρηματιστηριακές. Σε ό,τι αφορά την φορολογική μας πολιτική, σας ανακοινώσαμε εκ των προτέρων τις ε, δεσμεύσεις του Total σε ό,τι αφορά τη φορολογία, ε, δηλαδή το tax policy που λέμε, που υπάρχει και στο, στην ιστοσελίδα μας, τη φορολογική μας πολιτική, δεν θέλω να μακρηγορήσω από αυτού. Αυτό που προκύπτει σαφώς, όπως τόνισα, είναι ότι η σχέση ανάμεσα στον τόπο όπου παράγουμε ε, τα κέρδη μας και που πληρώνουμε τους φόρους είναι σαφέστατος ό,τι αφορά τις δραστηριότητε μας και η φορολογική ε, βελτιστοποίηση βραχυπρόθεσμα δεν είναι τμήμα των πρακτικών μας γιατί όταν η Total επενδύει σε μια χώρα, επενδύει για πολλά χρόνια ε, οι άδειε οι πετρελαϊκές ε, κρατάνε 20 με 50 χρόνια κατά μέσο όρο και είναι πολύ σημαντικό για μας να γίνουμε αποδεκτοί και να ε, φτιάξουμε σχέση εμπιστοσύνης με τα κράτη και με τις τοπικές κοινότητες με τις οποίες ε, συνεργαζόμαστε. Ε, το να πληρώσουμε αυτό που λέγεται το δίκαιο μερίδιο ας πούμε, φόρου στις χώρες όπου δουλεύουμε είναι τμήμα της, της πολιτικής μας για να γίνουμε αποδεκτοί. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι θα κάνουμε μια επιθετική φορολογική πολιτική και με μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα κέρδη, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί θα έχει μακροπρόθεσμα πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας. Για να τελειώσω, θα μιλήσω γρήγορα για τις φορολογικές συμφωνίες που ενδιαφέρουν κυρίως την Επιτροπή σας, ε, που έχουν μια τρομερή φήμη ε, μετά τα λεγόμενα LuxLeaks. Ε, οι συμφωνίες αυτές δεν είναι ένας τρόπος για να δοθούν πλεονεκτήματα που δεν πρέπει ε, σε ιδιώτες ή σε εταιρείε. Αντίθετα, τα ruling αυτά είναι ένα εργαλείο νομικής ασφάλειας για τις εταιρείε και για τα κράτη, γιατί επιτρέπουν στα κράτη να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείε ε, πληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις με, όπως καθορίζονται μέσω της νομοθεσίας. Δεν έχουμε κανένα ruling το το οποίο μας δίνει πλεονεκτήματα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και να επισύρει στρέβλωση του ανταγωνισμού και μια και δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν είμαστε αντίθετοι. Αντίθετα, είμαστε υπέρ της ιδέας ε, τα ruling να αποτελούν αντικείμενο πληροφόρησης και να υπάρχει ενημέρωση των φορολογικών αρχών. Δεν πιστεύουμε όμως αυτό το έγγραφο θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί, γιατί αν θέλουμε να εφαρμόσουμε... Ε, πρέπει να σας πω ότι μάλλον στην περίπτωση των ruling έχουμε πάρα πολλές ε, πληροφορίες για τις δραστηριότητε, για τα στοιχεία ενεργητικού που αν δημοσιευθούν θα δημιουργήσουν όντω προβλήματα ανταγωνισμού. Ε, δηλαδή μπορούν να πάνε στις φορολογικές αρχές αλλά όχι γενικά να δημοσιοποιηθούν. Ε, αυτά ήταν κάποια πρώτα λόγια γενικά και μετά είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως να σας πω ε, για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σίγουρα θα ακουστούν πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Μάρτιν Μακιούν που είναι επικεφαλής φορολογικών υποθέσεων της εταιρείας SSE. Καλημέρα, ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να σας απευθύνω το λόγο σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερω που μπορώ να παρίσταμαι εδώ στι εργασίε τη Επιτροπή για το πολύ σημαντικό θέμα τη φορολογική διαφάνεια. Είμαι, ονομάζομαι Μάρτιν Μοκίων και είμαι επικεφαλή ε, φορολογική υπηρεσία τη ΕΣΕΣΥ, μια ενεργειακή εταιρεία συγμένη στο Βρετανικό Χρηματιστήριο που δραστηριοποιείται στι αγορέ ενέργεια του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ιρλανδία. Δεν είμαι στη θέση να εξετάσω το συζήτημα των tax rulings ή αντίστοιχων μέτρων σε διάφορε επικράτε, γιατί η εταιρεία μου δεν τα έχει αξιοποιήσει ποτέ. Όμω μπορώ να σα μιλήσω για την πρόσφατη εμπειρία τη SSE για την βελτίωση τη φορολογική διαφάνεια και πιο συγκεκριμένα την διαδικασία που περάσαμε για να λάβουμε το πιστοποιητικό του Fair Tax Mark. Θα σα παρουσιάσω σύντομα την εμπειρία μα, γιατί επιλέξαμε αυτή την οδό και γιατί θεωρούμε ότι η ανεξάρτητη πιστοποίηση είναι τόσο σημαντική. Αν έχετε πιο τεχνικά ερωτήματα, βεβαίω να σα ε, απαντήσω στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των απαντήσεων. Αρχικά, τι είναι αυτό το ε, σήμα δίκαιων φόρων. Είναι ένα ανεξάρτητο πιστοποιητικό που είναι διαθέσιμο στο Μήνο Βασίλειο για καταναλωτέ και άλλα ενδιαφέρουσα μέρη, για ούτως ώστε, μάλλον ούτω ώστε οι καταναλωτέ και άλλα μέρη να εμπιστεύονται ε, ότι οι, τις και ότι έχουν καταβάλει δίκαιου φόρου. Τι σημαίνει όμω πραγματικά δίκαιο ουσιαστικά η αντίληψη ότι μια επιχείρηση ε, καταβάλει ένα δίκαιο επίπεδο και συντελεστή φόρων επί των κερδών της στην κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος. Δηλαδή δεν είναι μία ποινή επί του ε, κέρδους, είναι ο τρόπος που οι εταιρείες μπορούν να επιστρέψουν κάτι στην ε, κοινωνία τους είναι, το Fair Tax Mark είναι μια σχετικά νέα πρωτοβουλία στο Βασίλειο που λαμβάνει νέα δυναμική, όμως ε, προς το παρόν είμαστε η μοναδική εταιρεία στο FTSE 100 που έχει ε, λάβει το πιστοποιητικό αυτό. Πρόσφατα αναθέσαμε στην YouGov ε, εταιρεία δημοσκοπήσεων μία έρευνα σε ό,τι αφορά το, την κοινή γνώμη είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα. Μόλις 34% της κοινή γνώμης θεωρεί ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, πληρώνουν ε, τους ε, φόρους που τους αναλογούν, ε, ενώ κατά το 80% θεωρούν ότι το καταβάλουν ε, τους φόρους σε μικρές επιχειρήσεις. Το 10% μόνο θεωρεί ότι είναι επιτρεπτό για μια επιχείρηση να μεταφέρει ε, την έδρα της για να αποφύγει τον εταιρικό φόρο και μόλις 6% θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις δίνουν ακριβή στοιχεία για τη φορολόγηση. Επομένως αυτά μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Γιατί δεν θέλουμε να πιστεύει ο κόσμος ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων προσπαθεί να παρακάμψει τους κανόνες προς όφελός της. Έχουμε ήδη δει πόσο σημαντική είναι η εταιρική φορολόγηση για την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και για την εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και μεγάλων επιχειρήσεων. Ε, ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μας όλη αυτή η εμπειρία, ε, με τα καλά και τα αρνητικά της στοιχεία. Τελικά όμως ε, λάβουμε το πιστοποιητικό, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια υπεύθυνη στάση απέναντι στη φορολόγηση και διαφανή. Εμείς δημοσιοποιήσαμε την φορολογική μας πολιτική και προέβημε και στην υποβολή εκθέσεων αναχώρα, και δημοσιοποιήσαμε όλα αυτά τα στοιχεία. Επίσης, ε, δημοσιοποιήσαμε πολύ περισσότερα στοιχεία για το φορολογικό μας άχθος και περαιτέρω εξηγήσει, ούτω ώστε όλοι να κατανοούν και τα κίνητρά μας. Τελικά, ακούσαμε ε, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν τα είχαμε ξανακούσει στο παρελθόν. Εκτεθήκαμε και στην εξωτερική εξέταση και αξιολόγηση και αντιλήσαμε μαθηματικά και διδάγματα. Είμαστε επίσης ε, ε, θετικά διακείμενοι στα βελτιωμένα πρότυπα που θέτει το ε, σήμα δίκαιο φορολόγησης. Και αυτό θεωρώ ότι μα βγήκε σε καλό. Σε ό,τι αφορά όλη τη διαδικασία, πράγματι ορισμένε κυβερνήσει αναλαμβάνουν δράση, όμω ένα τομέα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να μα βοηθήσουν για να μάθει και η κοινή γνώμη τι συμβαίνει. Ε, τέτοιες κινήσεις όπως είναι το BEPS του ΩΣΑ ε, Επίση, έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε ό,τι αφορά την φορολογική δικαιοσύνη. Αλλά από τη δική μα κοπιά θεωρούμε ότι και οι επιχειρήσει πρέπει να αναλάβουν σημαντικό ρόλο ε, με το να είναι υπεύθυνε και διαφανεί. Γι' αυτό κάναμε και ό,τι κάναμε εμεί. Η προσέγγιση μα μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλου. Όμω θεωρούμε ότι ο καλύτερο τρόπο να χειριστούμε αυτά τα ζητήματα είναι να ακούσουμε πραγματικά τι έχουν να πούν οι καταναλωτέ, ε, οι πελάτε μα δηλαδή και η κοινή γνώμη και να είμαστε να τον πιο διαφανεί και ανοιχτοί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μακιόν. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κριστιαν Κομολετιμό που είναι αρμόδιος για φορολογικά θέματα στον όμιλο BNP Paribas. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ως Ευρωπαϊκή Τράπεζα σημαντικότατο επίπεδου χαιρόμεθα που μπορούμε να συμμετάσχουμε στις εργασίες σας και έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για την ε, δική μας εμπειρία. Αν επιτρέπετε να πω τι ρόλο παίζουμε στην οικονομία. Σήμερα η BNP Paribas είναι παρούσα σε 75 χώρες. Έχει 180.000 συνεργάτες από 150 χώρες. Ένα μεγάλο τμήμα είναι στη Γαλλία, 48% στις άλλες χώρες και 21% στον υπόλοιπο κόσμο. Το μεγαλύτερο λοιπόν τμήμα των δραστηριοτήτων μας είναι στην Ευρώπη. Ο όμιλός μας έχει δύο μεγάλους πόλους δραστηριοτήτων. Από τη μία η Τράπεζα Ιλιανικών Υπηρεσιών, δηλαδή ε, έχουμε ένα δίκτυο από ειδικέ τράπεζες ε, για να χρηματοδοτούν ε, για παράδειγμα τις επιχειρήσεις ή τον ασφαλιστικό και έχουμε και την επενδυτική τράπεζα οι βασικέ μας είναι οι τράπεζε για τι ε, τρέχουσες ε, τραπεζικές υπηρεσίε, Οι άλλε δραστηριότητε είναι μόνο 27%. Το BNP Paribas είναι η πρώτη τράπεζα στην Ευρώπη από πλευρά επιχειρήσεων και ε, πελατών και εξυπηρετούμε πάνω από 20 εκατομμύρια διαφορετικούς πελάτες. Εξυπηρετούμε λοιπόν. Πώς εργαζόμεθα λοιπόν Εργαζόμεθα, όπως περισσότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, υποκείμεθα λοιπόν σε φορολογικούς ε, κανόνες. Για να συνοψίσω. Ο όμιλός μας, όπως κάθε παρόμοιος όμιλος, θέλει να είναι απόλυτα νομοταγής. Και κάνουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε απόλυτα νομοταγής ε, όσον αφορά τη φορολογία. Θέλουμε να σεβόμεθα όλους τους κανόνες στα κράτη στα οποία λειτουργούμε και κάνοντας αυτό Θέλουμε σε κάθε κράτος όπου έχουμε δραστηριότητα να λαμβάνει τους φόρους που πραγματικά πρέπει να λαμβάνει. Προσπαθούμε λοιπόν να συμμορφωνόμαστε και να σας δώσω μερικά στοιχεία για τους φόρους που, ε, που πληρώνουμε πριν μιλήσω για τους κανόνες. Φόροι τώρα που πλήρωσε ο Όμιλος στη Γαλλία το 2014. Όλοι οι φόροι μαζί είναι 2,2 δις. Ποιο είναι το ενοποιημένο αποτέλεσμα, 3,9 δις. Δηλαδή 56% και μισό είναι ο φόρος που πληρώνουμε επί των κερδών. Αυτά τα 2,2 ε, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Ε, τα μισά περίπου είναι οι συγκεκριμένοι φόροι για τους συγκεκριμένους ε, τραπεζικούς και χρηματοδοτικούς τομείς, συστημικοί φόροι που είναι πολύ διαφορετικοί, αλλά και ο ΦΠΑ, που όπως ξέρετε στον τραπεζικό τομέα είναι πολύ συγκεκριμένος φόρος ε, και το πληρώνημα η επιχείρηση ενό άλλου τομείς μπορεί να μεταφερθεί στους ε, καταναλωτές. Εμείς πρέπει να πληρώσουμε λοιπόν το ΦΠΑ και επιπλέον στη Γαλλία η πληρωμή του ΦΠΑ συνοδεύεται με την πληρωμή του φόρου επί των ε, μισθών. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πρώτος φόρος. Ένα τέταρτο πάνω κάτω είναι ο εταιρικός φόρος και το υπόλοιπο είναι η λυπή. Τώρα να εστιάσω στο φόρο επί των εταιριών, τον εταιρικό φόρο, που είναι ο στόχος και των εργασιών σας. Ποια είναι η κατάσταση παγκόσμια, Συνολικά λοιπόν για τη δραστηριότητα του ομίλου μας, όχι μόνο στη Γαλλία, διαπιστώνουμε ότι ο φόρος που πληρώνουμε είναι 2,6 δις ευρώ επί ενός αποτελέσματος 3,1. Συνολικά λοιπόν ο εταιρικός φόρος είναι 85%, 85,4% των κερδών. Είναι αρκετά υψηλό. Αν εξαιρέσουμε τις χώρες όπου δεν είχαμε κέρδη, για να επικεντρωθούμε και να συγκρίνουμε τις χώρες όπου είχαμε κέρδη σε σχέση με το ποσοστό εταιρικού φόρου που πληρώσαμε, θα διαπιστώσουμε ότι αυτός ο συντελεστής δεν είναι τόσο ψηλός, δεν φτάνει το 80%, αλλά ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 28%, και κατανέμεται αρκετά ισότιμα ε, στο εσωτερικό των περιφερειών, 29-30% στα πλαίσια της Ένωσης ή της ευρύτερης Ευρώπης, 23% στην Ασία και την Αμερικανική Ήπειρο και την ε, ενώ η Αφρική και η Μέση Ανατολή είναι ανάμεσα με 26-27%. Αυτό το σημαντικό ποσό Πώς προκύπτει. Πρώτα απ' όλα διότι κυρίως τα δραστηριότητά μας είναι σε χώρες υψηλής φορολογίας. Κατά συνέπεια, βλέξτε, στη Γαλλία που είναι η έδρα μας και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ υψηλούς εταιρικούς, ε, φόρους, 38%, αλλά έχουμε μεγάλη παρουσία και στην Ιταλία και, και το Βέλγιο, όπου έχουμε 34 και 31,4 αντίστοιχα. Έχουμε ουσιώδη ρόλο στι ΗΠΑ όπου το ποσοστό εταιρικού φόρου είναι από 25% έως και 45% αν προσθέσουμε και τους πολιτιακούς εταιρικούς φόρους. Στη άλλη χώρη όπου ε, δραστηριοποιούμεθα είναι 30% για παράδειγμα και παραπάνω στη Βραζιλία, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Αυστραλία, μερικά μόνο παραδείγματα. Σε κάθε μία από αυτές τις χώρες Έχουμε μια πολιτική απόλυτη συμμόρφωση προς τη φορολογική νομοθεσία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σεβαστούμε απόλυτα τους ε, κανόνες και έχουμε επισημοποιήσει αυτή μας την πολιτική ε, εδώ και πολύ καιρό και αν εξετάσουμε τις χώρες όπου είναι χαμηλότερο το ποσοστό εταιρική φορολόγησης όπου δραστηριοποιούμε. Θα υπάρχουν μερικέ, διότι προσπαθούμε να βοηθούμε παντό του πελάτε μα παντού όπου έχουν ανάγκη ε, πιστώσεων, για παράδειγμα πιστώσεων εξαγωγικών. Αν εξετάσουμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση, υπό το φως των εκθέσεων ε, αναχώρα που αναφέρατε προηγουμένως κύριε Πρόεδρε, θα διαπιστώσουμε ότι οι χειρότερες επιδόσεις μας είναι εκεί που είναι πιο χαμηλή η φορολογία. Αυτό λοιπόν ε, αντιβαίνει τη συνήθη ιδέα ότι εκεί που είναι χαμηλή η φορολόγηση πάει κανείς για να επιτύχει κέρδη. Τουλάχιστον ο δικός μας όμιλος δεν έχει τέτοια πολιτική, όπως θα δείτε από τις εκθέσεις αναχώρα που δημοσιεύονται ε, ετησίω, θα σας επιτρέψουν να εξακριβώσετε ότι ούτως έχει κατάσταση. Προσθέτω επίσης ότι αυτές οι χώρες ε, χαμηλής εταιρικής φορολόγησης που πολλές φορές ε, θεωρείται ότι δεν συνεργάζονται, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια στις χώρες αυτές, εφόσον έχουμε δραστηριότητα, να υιοθετήσουν τις διεθνείς προδιαγραφές διαφάνειας και ανταλλαγής προφοριών. Έτσι λοιπόν ε, ο Παναμάς, όπου ε, δεν υπήρχε καλή συνεργασία, άλλαξε την ε, πολιτική του, ενώ για τις ε, Βρετανικές ε, Παρθένους νήσους, επειδή δεν είχαν σωστή συμπεριφορά, κλείσαμε την επιχείρησή μας εκεί. Δεν αντάλλασαν πληροφορία, δεν υπήρχε διαφάνεια. Πέρα από το σεβασμό των εθνικών κανόνων σε όλες τις χώρες όπου εργαζόμεθα, σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας συμμόρφωσης είναι η πολιτική τιμών μεταβίβασης. Ε, οι πολιτικές τιμών μεταβίβασης πολλές φορές έχουν κακή φήμη γιατί θεωρείται μεταφορά κερδών, αλλά στην πραγματικότητα είναι κανόνες που έχει ορίσει όσα που στοχεύουν να επιτύχουν την ε, αθέμητη μεταφορά κερδών και να διασφαλίσουν ότι τα κέρδη μένουν και φορολογούνται εκεί που ε, γίνονται. Έχουμε λοιπόν μια πολιτική και είμαστε μία από τους πρώτους ομίλους που υιοθέτησε μια πολιτική συνολικών και συνεπών τιμών μεταβίβασης παγκόσμια, εφαρμόζοντας πλήρως τις αρχές που καθόρισε ο ΩΣΑ και όπως είπα και προηγουμένως στοχεύουν κάθε κράτος να είναι κύριο του φόρου που του αναλογεί δηλαδή να αμείβεται το κράτος για τη δημιουργία αξιών στο έδαφος του. Αυτό είναι ο κανόνας που εφαρμόζουμε και η άλλη αρχή των τιμών ε, μεταβίβασης είναι να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση. Δηλαδή υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των κρατών για να αποφασιστεί ποιο τμήμα των κερδών πρέπει να φορολογηθεί σε ποια χώρα. Από αυτή την άποψη ο τραπεζικός τομέας σίγουρα δεν έχει τις δυσχέρειες που αναφέρθηκαν πρόσφατα σε άλλους τομείς και συμφωνώ με αυτό που είπε η συνάδελφός μου για το ότι έχουμε τη βάση μας σε κάθε χώρα. Η δραστηριότητά μας είναι πολύ κοντά στους πελάτες μας σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, δεν αξιοποιούμε τραπεζικές άδειες, άρα δεν υπάρχει ενδεχόμενο φυγής πόρων από τη μία χώρα στην άλλη για λόγους της λεγόμενης βελτιστοποίησης. Οι αρχές του ΟΣΑ στον τραπεζικό τομέα είναι ήδη πιο προωθημένες από τις αρχές σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, οι κανόνες ε, διανομής των κερδών που προσπαθεί να προωθήσει ο ΩΣΑ στα πλαίσια του ΜΠΕΠΣ εφαρμόζονται στον τραπεζικό τομέα. Αυτή η πολιτική λοιπόν των τιμών μεταβίβασης ελέγχεται συνέχεια τα τελευταία χρόνια από το σύνολο των ε, ε, φορολογικών αρχών σε όλες τις χώρες που εργαζόμεθα και όλοι λένε ότι είναι σύμφωνες με τις διεθνείς αρχές, ότι εφαρμόζονται με συνέπεια και συνέχεια, είτε έχουμε δηλαδή κέρδη είτε ζημίες και μας ε, διαβεβαίωσαν ότι έτσι το κάθε κράτος λαμβάνει το φόρο που δικαίως το αναλογεί. Για να καταλήξω σε αυτή την εισαγωγή μου, Είμαστε και σε χώρε με υψηλή εταιρική φορολόγηση. Δεν θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα αυτό. Θέλουμε να σεβόμεθα πλήρως και φροντίζουμε να σεβόμεθα πλήρως την ομοθεσία των κρατών αυτών. Και αυτή η συμπεριφορά αναγνωρίζεται και από τις εταιρείε κοινωνική αξιολόγηση που ανέφερα ο συνάδελφό μου προηγουμένω. που θεωρούν ότι η συμπεριφορά του BNP από πλευρά ε, φορολογική είναι απόλυτα υποδειγματική. Και φυσικά θα θέλαμε να υπάρξουν απλουστεύσεις που αναφέρεται όπως η εναρμόνιση του εταιρικού φόρου και μπορώ να επανέλθω αν υπάρξουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους τρεις. Πάμε στο, στις ερωτήσεις και απαντήσεις τώρα. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στην, στους δύο συνεισηγητές και καταρχάς στην Ελίζα Φερέιρα. Θα θέσω τις ερωτήσεις μου στα αγγλικά. Για ευκολία. Ευχαριστώ που ήρθατε και οι τρεις. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που μας διαμηνήσατε. Και ευχαριστούμε που είσαστε και διαθέσιμοι για να μιλήσετε με το Κοινοβούλιο. Που από μόνο του είναι απόδειξη της αναγνώρισης του, αναγνώρι... του γεγονότος ότι και οι εταιρείε έχουν το δικαίωμα ή μάλλον συγγνώμη, την υποχρέωση να εξηγήσουν ε, και στην κοινωνία τι κάνουν και όχι μόνο στους μετόχους τους. Ας μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα και σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας και τους τρεις σας το εξή. Όλοι δείχνετε να καταλαβαίνετε πως η εταιρική ευθύνη υπάρχει. Από την άλλη, έχουμε απέναντί μας πολλές εταιρείε που λένε ότι ο ανταγωνισμός είναι αμήλικτος και δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιου τύπου φορολογική συμπεριφορά εάν δεν το κάνουν και οι υπόλοιποι. Αυτό μας δεν έχει τελειωμό. Γιατί ο κόσμος χρειάζεται χρόνο για να αλλάξει. Και οι σημαντικοί παίχτες όπως οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να είναι ε, θετικό στοιχείο αλλαγής και όχι στοιχείο έτσι ε, χρονοτριβής ε, και καθυστέρησης. Αλλά τώρα πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να καταλάβω πώς αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας απέναντι στους άλλους ανταγωνές, ανταγωνιστές. Ε, δουλεύετε σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές ή ολιγοπολιακές αγορές. Οι δημοσιοποιημένες σας αυτές πρακτικές θεωρείτε ότι είναι πλεονέκτημα στις αγορές. Οι υπόλοιποι πώς βλέπουν αυτές τις πρακτικές, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζετε, που έχετε. Καθαρά οικονομικά. Ακόμα και αν από τη σκοπιά της ε, κοινωνίας αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε σίγουρα σε μια τέτοια έτσι, πιο υπεύθυνη φορολογική συμπεριφορά. Τώρα, ακόμα πιο λεπτόμερος. επί των παρουσιάσεων που κάνατε. Στην περίπτωση της BNP Paribas, διαβάσαμε στον τύπο ότι έχετε πάνω από 200 υποκαταστήματα σε φορολογικούς παραδείσους, όπως λέμε. Σωστό είναι αυτό. Άλλαξε. Ακόμα και αν μας λέτε ότι έχετε αυστηρό κώδικα διοντολογίας και συμπεριφοράς. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα παρόλα αυτά. Αναφέρατε τον Παναμά, ότι φύγατε από εκεί. Πώς καθορίζετε τι είναι φορολογικός παράδεισος. Είναι με βάση τον κατάλογο του ΩΣΑ, γίνεται αυτή η ερμηνεία ή έχετε και άλλα στοιχεία, μυστικότητα, ή χαμηλού φορολογικού συντελεστέ σε αυτές τις περιοχές. Έχετε αντίστοιχες πρακτικές απέναντι στους πελάτες σας, γιατί υπάρχει και πληροφορίες, υπάρχουν πληροφορίε, ότι οι περισσότερες τράπεζες βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν να καταβάλουν τους ε, φόρους τους. Όχι μόνο δηλαδή, δεν είναι το θέμα μόνο οι τράπεζες, αλλά και τι δραστηριότητες ε, ασκούν. Είναι, μια τέτοια, είναι τέτοια αυτή, έχετε αυτή την πρακτική. Λοιπόν εσείς, να βοηθάτε τους πελάτες σας. Στην περίπτωση της Total, είναι μια μεγάλη πολυεθνική η Total. Δεν έχετε φορολογική, επιθετική πολιτική και δεν, δεν προσπαθεί να κάνει τη λεγόμενη βελτιστοποίηση. Και υπάρχουν πολλοί Μερικέ φορέ πολύ χαμηλοί φορολογικοί συντελεστέ. Τι άποψη έχετε για αυτούς. Επίσης διαβάσαμε ότι το ΤΑΛ δημοσίευσε φέτος, αποφάσισαν δημοσίευση φέτος, το συνολικό αριθμό των ε, θηγατρικών τη. Αλλά είχαμε διαφορετικέ πληροφορίε. Ότι είχατε 30 ε, στην Ορλανδία, αλλά αυτό δεν κολλάει με άλλες ε, πληροφορίες που δόθηκαν για το, πάλι την Ολλανδία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να βρίσκεσαι στην Ολλανδία, ας πούμε. Είναι η δυνατότητα να μην φορολογούνται, ας πούμε, κάποια κέρδη ή τη δυνατότητα να μεταφέρεστε σε άλλες ε, χώρες. Θα κλείσετε επίσης εννέα ε, θηγατρικές στις Βαχάμες, στη Βερμούδα και στα νησιά Κέιμαν, σε τρεις φορολογικούς παραδείσους. Αναφέρατε αυτές σε νέα θηγατρικές, αλλά έχετε όμως 19 ακόμα θηγατρικές σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Είναι μια διαδικασία που είναι εξελίξη αυτή. Σε τι φάση βρίσκεστε. Τελικά ποια είναι τα σωστά νούμερα και ποια είναι η πραγματική στρατηγική. Και γιατί θεωρείτε ότι μόνο αυτές οι τρεις χώρες θεωρούνται φορολογική παράδειση. Γιατί εμείς, ε, υπάρχει ένα δίκτυο που έχει εντοπίσει 82 φορολογικούς παραδείσους. Έχουμε λοιπόν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες γύρω από το θέμα. Αναφέρατε πόσα μας δηλώνεται σε ό,τι αφορά το φορολογητέο εισόδημα, πόσα δηλώνεται στη Γαλλία, η διανομή που κάνετε παγκόσμια έχει κάποιο pattern που ακολουθεί. Και αν ναι, έχετε κάποια κέρδη που δεν δηλώνετε σε ορισμένες δικαιοδοσίες, σε ορισμένες χώρες. Είσαστε απόλυτα διαφανείς για την SSC. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό το βραβείο δημοσιοποιήθηκε αυτές οι άδειες που πήρατε, εν τόσο. Επίσης, είσαστε υπέρ των ε, καταχώρα εκθέσεων και υπέρ της απόλυτης διαφάνειας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του πράγματος. Μήπως ε, σας ζητάνε υπερβολικά πολλές πληροφορίες και αν υπερβολικά πολλές πληροφορίες μπορεί να θέσουν αμφιβόλο την ανταγωνιστική σας θέση απέναντι στους ε, άλλους ανταγωνιστές σας. και πόσο μακριά μπορούμε να πάμε στη διαφάνεια. Ούτω ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για σας στις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα να ανταποκριθείτε στις ε, ερωτήσεις των ε, πολιτών και των φορολογούμενων και στην ανάγκη για ενημέρωσή τους. Ο άλλος ε, συνεισηγητής, ο Μίκαλ Τόιερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, του κόσμου των επιχειρήσεων για την ε, επιθυμία τους και τη θέλησή τους να έρθουν εδώ και να τα συζητήσουν όλα αυτά μαζί μας. Εμείς ως ε, συνεισηγητές έχουμε πολλά ερωτήματα. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η Επιτροπή προσκάλεσε και άλλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που αρνήθηκαν να παρευρεθούν. Δεν μας ευχαριστεί βεβαίως αυτό. Ήθελα να το πω αυτό εισαγωγικά γιατί πολλές φορές δεχόμαστε πιέσεις όταν εξετάζουμε νομοθετικές προτάσεις. Τώρα εμείς έχουμε ερωτήσεις και επομένως σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπορούμε και εμείς να σας υποβάλουμε κάποια ερωτήματα για να κατανοήσουμε καλύτερα Ε, το σκεπτικό που ακολουθούν οι πολυθυμικές επιχειρήσεις ό,τι αφορά το φορολογικό του σχεδιασμό. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου προς εσάς. Για την Total πρώτα. Που αφορά την, ασχολείται μάλλον, δραστηριοποιείται στην πραγματική οικονομία και τα εμπορικά αγαθά. Επομένω θα ήταν πιο εύκολο κανείς ε, ε, να διερευνήσει και να αποδείξει την οικονομική ουσία. Αυτό θα ήταν πιο δύσκολο όταν πάμε στα χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά, όπου είναι πιο άειλα τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το φορολογικό σχεδιασμό, εξετάζεται επενδυτικά προγράμματα, όταν εξετάζεται το άνοιγμα νέων αγορών, ή τη μόνιμη εκπροσώπηση σας κάπου. Σίγουρα, πρώτα απ' όλα, θα διερευνήσετε τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν και ευκαιρίες που υπάρχουν στην νέα αγορά, στην οποία εισέρχεστε. Όμως, μετά υπάρχει και μεταγενέστερη συζήτηση και ανάλυση για τις φορολογικές επιπτώσεις. Και όλο αυτό ε, συμπεριλαμβάνεται στους επενδυτικούς υπολογισμού αν θέλετε, τη επιχειρησή σας. Μπορείτε να μα εξηγήσετε πώς γίνεται αυτό ακριβώς εσά. Μετά, κάτι το οποίο ανέφερε η συνάδελφος Φερέιρα, ε, οι εκθέσεις αναχώρα. Ξέρετε, το, πρόγραμμα BEPS του προτείνει τέτοιου είδους εκθέσεις αναχώρα προς τις φορολογικές ε, αρχές. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και οι επιστήμονες μας συνιστούν να εισαχθεί μια τέτοια υποχρέωση έκθεση αναχώρα στις ε, υποχρεώσεις ε, δημόσιων εκθέσεων. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα μπορούσε να αποκαλύψει επιχειρηματικά μυστικά και θα ήταν ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα για μια, για μια πολυεθνική ας που έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς έχετε μια θέση επί του ζητήματος αυτού. Τη δημοσίευση δηλαδή των εκθέσεων αναχώρα. Και τρίτον, θα ήθελα να θίξω το εξή. Α, το έχασα, θα επανέλθω στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από πλευρά του ΕΛΚ, η Ντανούτα Ευχαριστώ. Θέλω να σας ρωτήσω για το CCCTB, γιατί το αναφέρατε. Είναι η κοινή βάση για τον ενοποιημένο εταιρικό φόρο. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ την εθνική φορολογία. Και κατάλαβα από την κυρία Μονιετή ότι η εταιρεία σας ότι κάθε εταιρεία σε κάθε χώρα χρησιμοποιεί τις ε, εθνικές τιμές και δεν χρησιμοποιείται το σύστημα τιμών μεταβίβασης. Τι θεωρείτε λοιπόν για την ενοποιημένη βάση εταιρικού φόρου. Το δέχεστε ή λόγω του, της δομής ε, της, ε, του ομίλου σας είστε κατά. Δεύτερον, σε περίπτωση αντιδικιών για το θέμα του φόρου παγκοσμίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ε, διεθνών συγκρούσεων και αντιδικιών για φορολογικά θέματα. Ποιο θα ήταν το καλύτερο σύστημα για την επίλυση αυτών των ε, διενέξεων για φορολογικά θέματα. Θεωρείτε ότι λειτουργεί καλά, ικανοποιητικά το παρόν σύστημα για την επίλυση αυτών των διενέξεων. Ή θα προτιμούσατε ένα δεσμευτικό σύστημα διαιτησίας επίλυσης διαφορών. Είναι σημαντικό θέμα για σας αυτό. Και τελευταίο, για θέματα διαφάνειας. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι. Η διαφάνεια είναι η τάση. Ακόμη και αν κάποια τμήματα της προσπάθειας BEPS του ΟΣΑ, της προσπάθειας δηλαδή αντιμετώπιση των προβλημάτων μετατόπισης κερδών και διάβρωσης προλογικής βάσης. Η ερώτησή μου θα σας φανεί ίσως λίγο περίεργη. Θεωρείτε ότι οι πολυεθνικές έχουν συνέστηση ήδη ότι υπάρχει αυτή η νέα τάση η οποία θα ενισχυθεί και δεν είναι απλώς αποτέλεσμα του LuxLeaks αυτό που συμβαίνει. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος ότι θα υπάρξουν πιο καινοτόμες προσπάθειες ε, ε, προφορολογικού σχεδιασμού και κατάχρηση του συστήματο. Δηλαδή ότι αυτοί που θέλουν να καταχραστούν το σύστημα, να κάνουν κακή χρήση του συστήματο, πάντα θα είναι ένα βήμα μπροστά από αυτού που προσπαθούν να του ε, πιάσουν στα πράσα. Ποια είναι η αντίποσή σα για το τι γίνεται παγκοσμίω για να ενισχυθεί η διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ντανούτα. από, τους, από το ECR. Πίρκο Χουάναν Εμείς πάντα ήμασταν υπέρ της αναγνώρισης ότι η φορολογική πολιτική είναι αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους και επομένως τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τα συστήματα φορολόγησης. Η ομάδα μου είναι υπέρ των εργασιών της Επιτροπής και των κρατών μελών για να προωθήσουν την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε όλα τα απαραίτητα διεθνή βήματα. Θα ήθελα τώρα να θέσω τα εξή ερωτήματα. Τα ευρωπαϊκά κράτη πώς μπορούν να πλουστεύσουν τα φορολογικά συστήματα, ούτως ώστε οι εταιρείε να παίζουν ισότιμα εντός της ε, ενίας αγοράς. Ποια αφορολογικά καθεστώτα είναι τα πιο επιζήμια και ασαφή για τις εταιρείε και δεν τους επιτρέπουν να ανταγωνιστούν, να αναπτυχθούν και να επενδύσουν στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Άλντε. Τόρβαλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όπως και τα σπαγγέτι western, ασχολούμαστε με, το καλό, με τον καλό, τον κακό και το άσχημο. Εσείς φαινομενικά φαίνεστε καλοί της υπόθεσης, της ταινία. Μία ερώτηση για τις δομές, γιατί έχουμε στοιχεία για διαφορετική οικονομική ανάπτυξη για τις μεγάλες και μικρές χώρες. Αν σε ενδιαφέρει θεωρία, υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο του Και αυτή η διαφορετική οικονομική ανάπτυξη επιτρέπει, τις, ε, αναγκάζει μάλλον τις ε, μικρές χώρες με την χειρότερη, τις χειρότερες οικονομικές συνθήκες να μπουν στην προσπάθεια επιθετικής φοροαποφυγής. Όταν κοιτάτε τι κάνουν οι εταιρείες σας, θα πρέπει να είστε σε θέση να καταλάβετε αν αυτή η θεωρία έχει βάση. Έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη λόγω των, της σημερινής κατάστασης της οικονομίας, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης. Ο Φάμπιο Ντομάζη. Δεν, το, ένα σπαγκέτι, σπαγκέτ, western σπαγκέτι ε, ποτέ δεν είναι καλό εάν δεν έχει και λίγο μπαμπούμ, λίγο, λίγους πυροβολισμούς προς την PNB Παριμπά. Με βάση ένα άρθρο από το Huffing Post, η Παριμπά ε, πρόσφατα ε, έδωσε συμβουλές ε, σε κάποιους επενδυτές από την Ουκρανία να αποφεύγουν τη φορολογία χρησιμοποιώντας κάποιες εταιρείες offshore. Το κάνετε σε αυτό, σε επιχειρήσεις σας. Είχατε κάποιες αρνητικές εμπειρίες με τις εκθέσεις αναχώρα. Γιατί ο τραπεζικός τομέας είναι ο πιο περίπλοκος σε ό,τι αφορά την κερδοφορία και τις μετοχές κτλ. τα λοιπά. Η Total για τη διαφάνεια. Γιατί δεν συμπεριλάβατε τις 30 θηγατρικές από τις 178 που βρίσκονται στην Ολλανδία στον κατάλογο των 903 που δημοσιεύσατε το Μάρτιο του 2015. Και για ποιους λόγους το κάνατε αυτό. Δεύτερον, όπως είπε και η Λίζα Φερέιρα, κλείσατε μόνο 9 από τις 19 θηγατρικές της Βερμούδα, Μπαχάμες και στα Κέιμαν. Και αυτά που κλείσατε, αυτέ τι ιατρικές, χρησιμοποιόταν για φοροαποφυγή στο παρελθόν και γιατί τι κλείσατε. Και τέλος, γιατί έχετε τόσε πολλές επιχειρήσεις με... στην Ολλανδία, τόσες πολλές ιατρικές. Όχι μόνο γιατί η Ολλανδία σας επέτρεψε να έχετε βιβλία σε δολάρια, δεν είναι μόνο η μόνη χώρα, και τι ποσοστό των κερδών σα περνάει από την Ολλανδία. Η Total δεν πλήρωσε ε, το 12, το 13 και το 14 φόρους στη Γαλλία, παρά ότι ε, το 2012 ε, είχε 58 ε, δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος το 12, 40,3 ε, το 13. Τώρα είπατε θα πληρώσετε φόρους. έχετε διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο. Γιατί θα πληρώσετε φόρους τώρα ενώ δεν πληρώσατε πριν. Εκτός αν υπήρχε εταιρική φόρο αποφυγή στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γερανόπουλο. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση προς την, στον εκπρόσωπο της Παρίμπα που φαίνεται ότι εκτός των άλλων ειδικεύεται και στις συμβουλές προς τρίτους. Στην Ελλάδα υπήρχε μια μεγάλη τράπεζα εξειδικευμένη στην αγροτική οικονομία, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μέσω δανείων προς τους αγρότες έχει υποθηκευμένη ολόκληρη την αγροτική γη της Ελλάδας. Πριν από λίγα χρόνια η Μπά ήταν ο σύμβουλος, συμβούλεψε την τότε ελληνική κυβέρνηση να μεταβιβάσει, γιατί ήταν κρατική η τράπεζα, να μεταβιβάσει το υγιές τμήμα της τράπεζας αυτής εντελώς δωρεάν σε άλλη ιδιωτική τράπεζα το δε μη υγιές τμήμα να περάσει σε καθάριση. Καταλαβαίνετε εδώ ότι πρόκειται περί ενός σκανδάλου που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο στην Ελλάδα, στην οποία σύμβουλος ήταν η Παριμπά. Δεύτερο ζήτημα. Όπως όλοι γνωρίζετε, δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση κοντεύει σε συμφωνία ε, με τους τρεις θεσμούς για το γνωστό πρόβλημα. Ένα από τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας είναι η υπερβολική επιβάρηση για μία ακόμη φορά των λαϊκών στρωμάτων με πραγματικά εξοντοτικούς φόρους. Και είναι πρόκληση να συζητάμε σήμερα το καθεστώς των εταιριών με βάση το οποίο μπορούν να ξεφεύγουν από φόρους τους οποίους με τη σειρά τους φορτώνονται σε εργαζόμενους, ανέργους, μικροεπαγγελματίες κτλ. Έχω ένα ερώτημα για το τι πιστεύουν ε, οι εκπρόσωποι των εταιριών. Αν δεν υπήρχε η συνθήκη της ελευθερίας της κίνησης κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τη συνθήκη του Μάστριχτ, θα είχαν αυτή τη δυνατότητα, τελειώνω, αυτή τη δυνατότητα της ε, ε αντιμετώπισης των φορολογικών του υποθέσεων με τόσο προνομιακό τρόπο. Και κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Έχουν κληθεί μεγάλες εταιρείε να απαντήσουν σε ερωτήματα. Πολλές δεν απάντησαν, πολλές δεν αρνήθηκαν. Επειδή όμως οι εταιρείε λειτουργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εκμεταλλεύονται το πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήθελα να ρωτήσω αν η Επιτροπή, αν το Προεδρείο σκέφτεται να εισηγηθεί κυρώσει για αυτές τις επιτροπές και ένα δεύτερο ερώτημα, γιατί δεν έχουν κληθεί από την Ελλάδα η εταιρεία Coca-Cola 3E, ε, μεγάλη εταιρεία με έδρα φορολογική του Λουξεμβούργο, και δεύτερον η εταιρεία Eldorado με έδρα φορολογική την Ολλανδία είναι η γνωστή εταιρεία που έχει ξεσηκώσει αντιδράσει χωρί να πληρώνει κανένα φόρο, και κυριολεκτικά καταστρέφει το περιβάλλον σε μια μεγάλη περιοχή τη Ελλάδα. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Θα τα εξετάσουμε στην πορεία. Γιατί και οι Έλληνε εφοπλιστέ δεν πληρώνουν φόρου. Να το δούμε και αυτό το θέμα. Ε, Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Αναγκόμε για του ε, σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήμουν εδώ προηγουμένως, Ήταν όμως η βοηθή μου και μου μετέφεραν τα όσα διαμήφθησαν. Σημειώνω ότι αναφέρθηκαν φορολογικοί συντελεστέ ή μάλλον ε, το 85% που έχουν καταβληθεί σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Πρέπει να έχετε καλύτερου συμβούλου τότε, αν ε, πληρώνετε τέτοιου φόρου. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Ποια θεωρείτε πρέπει να είναι η δημόσια πολιτική σε ό,τι αφορά την δίκαιη φορολόγηση. με βάση και τα όσα προτείνονται από τον Επίτροπο Μοσκοβισή, η πρόταση που δημοσιεύτηκε, ποια είναι η γνώμη σας απέναντι στα μέτρα που προτείνει για την αποφυγή της μεταβίβασης ε, τιμών μέσω και του CCTV και ποια είναι η θέση σας σε ό,τι αφορά την έκθεση αναχώρα και για την υποχρέωση ε, τέτοιων εκθέσεων. Παρακαλώ κύριος Μόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προ την ΠΕΝ Παριμπά θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημά μου. Ποιο είναι ο κύριο ε, λόγο ε, που εγκαταστήσατε την εταιρεία σα στο Λουξεμβούργο εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά ε, τι είδους ε, φορολογική συμφωνία έχει συναυθεί για κατά τη διάρκεια όλης αυτής της ε, κατάστασης και ποια είναι η σύγκριση με την φορολόγηση εκτός καθεστώτος tax ruling που θα μπορούσε να είχατε καταβάλει τότε. Από το EFTD δεν έχω λάβει αίτημα δεν θέλει κάποιος να μιλήσει, να μιλήσει δηλαδή να πάρει το λόγο. Να ξαναδώσουμε το λόγο λοιπόν στους ομιλητές μας. Θα ξεκινήσουμε από την ΠΕΝΠΕ, μετά SSC και μετά το ΤΑΛ. Παρακαλώ κύριος Κομολέ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι ακούστηκαν πολλά ερωτήματα. Ελπίζω να μην παραλείψω τίποτα. Ένα πρώτο ερώτημα αφορούσε την παρουσία μας στους φορολογικούς παραδείσους. και αναφερθήκατε σε συγκεκριμένε μελέτες μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. Υπάρχει έλλειψη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά τα λογιστικά στοιχεία και έτσι χάνουν και το δίκιο τους εν μέρη. Αφενός είναι απαράδεκτο να εξετάζουμε τον ίδιο τρόπο τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική δραστηριότητα, δηλαδή εκατοντάδες ή χιλιάδες εργαζόμενοι που ισχύει για μας, με άλλες περιπτώσεις όπου έχουμε απλώς ε, χρηματοοικονομικές ροές που διέρχονται από μια συγκεκριμένη επικράτη. Αυτό είναι η πρώτη αδυναμία. Δεύτερη αδυναμία. Αυτοί οι κατάλογοι συχνά γίνονται έτσι αυτοσχέδια ή με πολύ παλιά στοιχεία της δεκαετίες του 70 και έτσι δεν λαμβάνουν ε, καθόλου υπόψη τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Τι συνέβη λοιπόν. Τον Οκτώβριο του 2008 είχαμε την πρώτη διεθνή διάσκεψη για τους φορολογικούς παραδείσους που είχε συνδιοργανωθεί από Γαλλία και Γερμανία. Στο G20 το Νοέμβριο του 2008 όταν τα ξανασυζητήσαμε όλα αυτά είχαν αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Θεσπίσαμε ένα παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια ε, υπό την αιγίδα του G20, του, του που είναι όμως πολύ ευρύτερο ε, πλαίσιο, με πολύ περισσότερα μέλη. Και σε σχέση με αυτόν τον κατάλογο κατατάσσονται και τα κράτη σε διάφορες κατηγορίες. Ότι συμμορφώνονται, δεν συμμορφώνονται ή συμμορφώνονται εν μέρη. Και με αντικειμενικότατο τρόπο, γιατί ξέρετε ότι πρέπει να γίνονται πολύ σοβαρά αυτές οι διεργασίες, με πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά πρότυπα, θεωρητική εξέταση και μετά και πρακτική εξέταση από ομοτήμους. Είναι λοιπόν ένα ιδιαίτερα αντικειμενικό πλαίσιο που ένας μεγάλος ε, όμιλος όπως ο δικός μας ε, παραπέμπει και αναφέρεται μάλλον και σε αυτόν τον κατάλογο. Αναφερόμαστε επίσης ε, σε άλλο κατάλογο της Γαλλίας που δημοσιεύεται ε, κάθε χρόνο από τη Γαλλία, θα σας έλεγα, αλλά σήμερα, 23 Ιουνίου, θα έπρεπε να έχει ήδη από την 1η Ιουνίου δημοσιευθεί αυτός ο κατάλογος. Αλλά τέλος πάντων, η αρχή υφίσταται. Αυτός ο γαλλικός κατάλογος που επικαιροποιείται λοιπόν κάθε χρόνο και ο διεθνής κατάλογος, ε, αποτέλεσμα επικοδομητικής συνεργασίας όλων αυτών των ε, μελών, σε όλα αυτά λοιπόν αναφερόμαστε. Συμμετέχουμε λοιπόν σε όλες αυτές τις διαδικασίες και σε ό,τι αφορά την φορολογική διαφάνεια. Έχουμε πραγματική δραστηριότητα. Αναφέρθηκε προηγουμένω το Λουξεμβούργο, αλλά έχουμε εκεί πέρα 3.500 μέλη προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της απόκτησης ε, της φόρτης, όταν εκεί εξαγοράσαμε τη φόρτης λοιπόν, η φόρτη είχε την τράπεζα BGL, που είναι η μεγαλύτερη τράπεζα του Λουξεμβούργου. Έχουμε πελατολόγιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή και ιδιωτών στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται λοιπόν για πραγματική δραστηριότητα. Και εξάλλου στι μελέτε των μη κοινωνικών οργανώσεων που αναφερθήκατε, υπάρχουν πολύ συχνά υποσημειώσει ότι ναι, δραστηριοποιούνται μεν ε, στο Λουξεμβούργο, αλλά υπάρχει πραγματική δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για ε, το Βέλγιο, που θεωρείται από μερικού ε, φορολογικό παράδεισο. Ε, για μας αυτό δεν έχει νόημα. Είμαστε η πρώτη τράπεζα στο Βέλγιο. Και ο εταιρικό φόρος είναι πάνω από 30%. Σε αυτές τις μελέτες λοιπόν είναι πολύ λανθασμένη η προσέγγιση. Εμείς ακολουθούμε τις αρχές αυτών των καταλόγων στους οποίους συμμετέχουμε. Μεριμνούμε για τη διαφάνεια στις χώρες όπου δραστηριοποιούμεθα και ακόμα και σε φορά τη πιο ελαφριά εντός φορολόγηση. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε διατάξεις στη Γαλλία, ούτως ώστε να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε οντότητε ε, όταν υπάρχει το, ένα, σε χώρες που υπάρχει αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο, γιατί θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το ελαφρύτερο φορολογικό πλαίσιο. Επομένως, το καθεστώς αυτό ε, που αξιοποιείται στο τοπικό επίπεδο δεν συνδέεται με το πιο ευνοϊκό συντελεστή που θα μπορούσε κάποιος να αξιοποιήσει ε, στη Γαλλία. Δεν το συγκρίνουμε δηλαδή με αυτό αλλά με τον κλασικό συνήθι συντελεστή. Αν δούμε τα τελευταία δέκα χρόνια, δεν υπήρξε περίπτωση που θα έπρεπε να γίνει επίκληση αυτής της διάταξης ό,τι αφορά την, ε, τον ομιλό μας. Επομένως, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ε, παρουσία μας ε, σε αυτέ τι χώρε με πιο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο. Μετά, τι συμβαίνει με τους πελάτε μας. Και εδώ είναι σαφή τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Οι τράπεζες και οι BNP και οι υπόλοιπε είναι ε, η πρώτη βοηθητική υπηρεσία, αν θέλετε, απέναντι ε, στις φορολογικές αρχές. Και στα χρηματοπιστωτικά μέσα και αγαθά, βοηθούμε τις φορολογικές αρχές, αλλά και ε, για να συλλεγούν δηλαδή οι φόροι, αλλά συλλέγουμε και πληροφορίες και στοιχεία για τις φορολογικέ αρχές. Κάνουμε λοιπόν αυτή την εργασία ε, με τη μορφή της ε, ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος και τώρα έχουμε περάσει σε μία νέα φάση με αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και με την οδηγία του 2005 με πολύ στενό όμως πεδίο εφαρμογής γιατί αφορούσε μόνο την αποταμίευση και με τις ΕΙΠΑ αλλά και με την αυτόματα τώρα ανταλλαγή πληροφοριών ε, στο πλαίσιο του ΩΣΑ αλλά και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο με την διεύρυνση ε, του φάσματος των ε, προϊόντων που καλύπτονται και κάθε φορά οι τράπεζες ε, ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόκληση, έκαναν και τις ε, τεχνικές και οικονομικές επενδύσεις για να ε, πληρούν και τα νέα κριτήρια. Εμείς λοιπόν επιτελούμε αυτό το έργο με ευσυνειδησία. Να προσθέσω εδώ ότι σε ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε είναι πιο ανεπτυγμένος ο ιδιωτικός ε, τραπεζικός κλάδο, ή μάλλον των ιδιωτών. Εμείς ε, αξιοποιούμε άλλες ε, δραστηριότητες και για αυτές είμαστε απόλυτα σαφείς και καθαροί με τις υποχρεώσεις μας. και αυτή τη φορά και τους πελάτες μας βεβαίως, πέραν των υποχρεώσή της τη μας της δημοσιονομικής. Έγινε μια ερώτηση για το εάν και κατά πόσο το θέμα της επίλυσης φορολογικών διενέξεων είναι θέμα. Έχετε δίκιο κυρία μου που το αναφέρετε. Τι διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια ο μηχανισμός ε, αποφυγής της διπλής επιβολής, της διπλής φορολόγησης που ήταν ε, βασικός ε, κανόνας των διεθνών φορολογικών ρυθμίσεων λειτουργεί όλο και χειρότερα. Και γιατί. Γιατί. Πρώτον, δεν καλύπτει όλους τους φόρους αυτός ο μηχανισμός. Επιπλέον, η έλεγχη είναι όλο και πιο συχνή και όλο και πιο πολύ σε βάθος και υπάρχουν και διαφορές ερμηνεών μεταξύ φορολογικών δικήσεων, άρα έχουμε όλο και περισσότερες περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, ακόμη και τριπλής και τετραπλής σε ορισμένες περιπτώσεις, για να το πούμε όλα. Οπότε, ορισμένες φορές ο μηχανισμός αυτός δεν λειτουργεί, γιατί επειδή κάπου έχει υπάρξει μια κύρωση, που δεν ξέρουμε αν τελικά όμως θα διατηρηθεί, θα γίνει τελεσίδικη, γι' αυτό ορισμένε ε, φορολογικές διοικήσεις αρνούνται το θέμα αυτό να εξεταστεί στα πλαίσια μιας ε, φιλικής επίλυσης διαφορών. Και ε, σε άλλες περιπτώσεις είναι τόσο ο φόρτος εργασιών των διοικήσεων, των εφοριών, έχουν τόσο πολλά θέματα που τραβάνε πολύ οι υποθέσεις αυτές. Οπότε το θέμα που τίθεται και που πρέπει να τονιστεί είναι δεν θα έπρεπε να αναπτύξουμε δεσμευτικούς, χρεωτικούς μηχανισμούς επίλυσης ε, διαφορών μεταξύ φορολογικών διοικήσεων. Πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί και στην Ευρώπη που έχουμε αυτή τη σύμβαση για τις διατησίες, για τις ε, τιμές ε, μεταβίβασης, θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής τους. Αλλά ούτως άλλως αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου δύο περιπτώσεις, ε, μία το τρία, μία το πέντε και τα τελευταία 10 χρόνια δεν θυμάμαι απ' έξω, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία περίπτωση. Μία-δύο. Άρα υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές περιπτώσεις διπλής φορολόγησης. Ποιος θα έπρεπε να είναι ο στόχος. Οι δημόσιες αρχές ε, να επιδεικνύουν συνέπεια. Δηλαδή, Βεβαίως να πολεμούμε την ε, φοροδιαφυγή, τη διάβρωση της φορολογικής βάσης, όλα αυτά είναι απαράδεκτα και μειώνουν τα κρατικά έσοδα. Αλλά παράλληλα πρέπει να φροντίζουμε οι επιχειρήσεις που είναι οι πιο νομοταγείς να μην αντιμετωπίζονται συστηματικά χειρότερα από τους άλλους και να μην πληρώνουν διπλά φόρο συστηματικά. Τώρα, τέθηκε ένα συγκεκριμένο θέμα για το Λουξεμβούργο. Και εδώ ήδη το ανέφερα. Έχουμε ουσιώδη πραγματική παρουσία. Είμαστε τράπεζα που λειτουργεί, δραστηριοποιείται επί τόπου. τώρα στο Λουξεμβούργο αλλά και σε άλλες χώρες ε, που εργαζόμεθα ζητήσαμε να υπάρξουν φορολογικές συμφωνίες αυτή τη στιγμή έχουν θετική, έχουν συγγνώμη, αρνητική ε, φήμη ε, ενώ είναι τόσο διαδεδομένες γιατί υπάρχουν σε 23 από τις 28 χώρες είναι καλή πρακτική αυτή των συμφωνιών είναι μια πρακτική την οποία έχει ενθαρρύνει το φόρουμ του ΟΣΑ για τις ε, φοριακές αρχές που δημιουργήθηκε το 2002 θεωρώ ότι είναι καλές αυτές οι πρακτικές. Αυτό τι σημαίνει για μια εφορία. Ότι υποχρεώνεται να λάβει θέση για να διευκρινιστεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι και ο φορολογούμενος έχει μια ασφάλεια. Μια ασφάλεια που είναι λογικό να την αναμένει. Άρα είναι πολύ καλή πρακτική. Ε, καλύτερα θα ήταν λοιπόν να επεκταθεί αυτή η πρακτική. Βέβαια δεν περιέχει κινδύνους. Βέβαια πάντα υπάρχουν κίνδυνοι. Ο κίνδυνος είναι ότι αντί να ερμηνεύσει τον νόμο η εφορία στην οποία υποβάλλεται το αίτημα απομακρύνεται από τον νόμο. Αυτό βέβαια δημιουργεί κίνδυνο. Είτε κρατικής επιδότησης, για παράδειγμα, αν αφορά μερικές επιχειρήσεις ε, τοπικές, είτε αθέμη του φορολογικού ανταγωνισμού, αναφορά επιχειρήσει που δεν έχουν την έδρα του εκεί, αλλά αυτό ο κίνδυνο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όχι. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Νομίζω έχουμε μία λύση θαυμάσια που την πρότεινε στι 18 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών συμφωνιών μεταξύ εφοριών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Σαφέστατο. Ο κύριος Μακιούεν. Thank um, Έχουμε δραστηριότητε ε, ουσιώδει σε δύο χώρε. Η θέση μα είναι κάπω λοιπόν διαφορετική από την BNP Paribas και Total που είναι πραγματικέ πολυεθνικέ. Ποια είναι η θέση η δική μας, SSE. Είμαστε μια εταιρεία που επιδιώκει μακροχρόνια βιωσιμότητα. Δεν θέτουμε το βραχυπρόθεσμο κέρδο σε αντιπαράθεση με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Όταν καθορίσαμε την φορολογική μας θέση, το συζητήσαμε με τους μετόχους, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς. Θέλουμε να είμαστε υπεύθυνη εταιρεία, υπεύθυνη επιχείρηση. Είδαμε και άλλες ε, εταιρείες που κάνουν δηλώσει ότι αυτές οι εξελίξεις μπορεί να έχουν επιπτώσεις ε, στα κέρδη μακροπρόθεσμα. Όμως εμείς ε, και οι μέτοχοί μας δεν θεωρούμε κάτι τέτοιο. Τι έχουμε κάνει λοιπόν για το φόρο. Οποτεδήποτε χρειάστηκε να το κάνουμε, το κάναμε εθελουσίως. Ακούσαμε δηλαδή τι μας λένε οι πελάτες μας και ακούσαμε και τι λέει και η ευρύτερη κοινή γνώμη. Τώρα για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που τέθηκαν. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για τους ανταγωνιστές μας, αλλά για το οικονομικό όφελος των ενεργειών μας για, αυξημένη διαφάνεια στα φορολογικά μας. Ήμασταν απόλυτα ανοιχτοί. Δεν χρησιμοποιούμε κανένα μηχανισμό φοροαποφυγής. Και αυτό νομίζω ότι μας δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διότι οι πελάτες μας θέλουν να συναλλάσσονται με καλές και υπεύθυνες εταιρείε. Και νομίζω ότι τελικά θα έχουμε μακροπρόθεσμο όφελος. Όπως είπα και προηγουμένως, εμείς ε, θελήσαμε να έχουμε από έναν εξωτερικό φορέα αυτό το σήμα ότι είμαστε υπεύθυνοι στα φορολογικά μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα αντιμετωπίσει πολύ θετικά αυτό. Θα παραλαμβάνω. Αυτό είναι βάση μια σειρά πρωτοβουλειών μας, ούτως ώστε να φαινόμεθα ότι λειτουργούμε με μακροπρόθεσμο, υπεύθυνο, βιώσιμο τρόπο όσον αφορά τη φορολόγησή μας ή και για άλλα θέματα. Τώρα για το θέμα των εκθέσεων αναχώρα. Εμείς το κάνουμε θελουσίως. Βέβαια είναι πολύ λιγότερες αυτές οι εκθέσεις αναχώρα από ότι οι εκθέσεις πρέπει να κάνει το Τάλκι Παριμπά ότι αυτοί δραστηριοποιούνται σε πολύ περισσότερες χώρες. Αλλά πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία ξέρετε. Πρέπει να δώσουμε επαρκή πληροφόρηση, ούτω ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλαβαίνουν ποια είναι η οικονομική μα δραστηριότητα, ποια είναι τα έσοδά μας, τα κέρδη μας και ο φόρος που πληρώνουμε στις διάφορες φορολογίες. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε εμπορικά εμπιστευτικές πληροφορίες. Πρέπει να δούμε δηλαδή ποια είναι η ουσία των πληροφοριών που δίνεις. Βεβαίως να δώσεις την πληροφορία που θα χρησιμοποιηθεί και που είναι χρήσιμη για τους άλλους. Τώρα για αυτό το θέμα CCCTB του ενιαίου εταιρικού φόρου. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ε, χωρών. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί οι κανόνες για τις τιμές μεταβίβασης και για την επίλυση διαφορών. Πρέπει να υπάρχει περισσότερο συντονισμός γι' αυτό μεταξύ των ε, φορολογικών αρχών των διαφόρων κρατών. Όσο περισσότερη τέτοια συνεργασία, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η φοροαποφυγή. Ανταλλαγή πληροφοριών. Απόλυτα στοιχείο κλειδί. Λοιπόν, εμείς ως SSE στηρίζουμε οτιδήποτε που θα αυξήσει τη διαφάνεια και τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ φορολογικών συστημάτων, ούτω ώστε να λειτουργούν, να εφαρμόζονται κανόνες και να πληρώνουν το δίκαιο και σωστό φόρο οι εταιρείε. Διότι ξέρετε, ο καθένας πρέπει να παίξει το σωστό του ρόλο για να επιτύχουμε σωστό και ισότιμο ε, ανταγωνισμό. Οι εταιρείε πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες, οι κυβερνήσεις πρέπει να καθορίζουν και να εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες και υπάρχει και το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΣΑ που έχουν κρίσιμο ρόλο να παίξουν για να επιτευχθεί ο συντονισμός. Αυτοί λοιπόν οι τρεις φορείς ο καθένας στο επίπεδό του Ελπίζουμε τουλάχιστον ότι θα μας βοηθήσουν σε ένα, για να επιτύχουμε ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα παγκοσμίω. Αλλαγές στις τιμές μεταβίβασης. Είναι θέμα κλειδί. Και πάλι, οι τιμές μεταβίβασης, οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι σημαντικό στοιχείο για να αποφευθεί η φόρο αποφυγή. Οι κανόνες λοιπόν αυτοί για τις τιμές μεταβίβασης πρέπει να είναι συντονισμένοι. Και η εργασία που έχει κάνει η ΩΣΑ και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να στηριχθούν οπωσδήποτε, ούτως ώστε αυτοί οι κανόνες να λειτουργούν σωστά όπως ήταν ο στόχος τους. Το αυτό για τις εκθέσεις αναχώρα. Αν πρέπει να είναι υποχρεωτικές. Δύο τρόπους έχουμε για να επιτύχουμε βελτίωση. Εφελούσια και υποχρεωτική υποβολή. Νομίζω ότι από τη μία θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνε οι εταιρείε και να δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τους. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά αν αυτό δεν επιτύχει το επίπεδο διαφάνειας που επιδιώκουμε, ούτω ώστε οι εταιρείε να καταλαβαίνουν και η κοινή γνώμη ότι πληρώνουν το σωστό φόρο, τότε το επόμενο βήμα το λογικό θα είναι υποχρέωση. Και νομίζω ότι ούτω ή άλλω ε, θα αξιοποιήσουμε αυτό το μέσο, την ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα, μεταξύ και άλλων μέτρων. Αυτά νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια εντάξει, εμείς ε, είμαστε σε διαφορετική θέση από τους άλλους δύο εδώ συνομιλητές μου. Σαφέστατο. Η κυρία Μονιετή, τελευταία. Ευχαριστώ. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω κάποιες και να απαντήσω σε ομάδες λοιπόν ερωτήσεων. Να απαντήσω στον αστεϊσμό, ότι είμαστε ανοργάνωτοι ε, αν πληρώνουμε εταιρικό φόρο 85%. Όχι, τόσο πληρώνουμε. 78% στην Νορβηγία, ε, λιγότερο στην Αφρική κτλ. Ε, έχει να κάνει με τις δραστηριότητές μας, ε, που είναι η αναζήτηση, η διερεύνηση για την ύπαρξη υδρογων ανθράκων. Ε, ο μέσος φορολογικός τελεστής είναι πάνω από 50% και αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η φορολογική... Ε, συγγνώμη, η πετρελαϊκοί αυτή η πόρη είναι πολύ σημαντική για τις χώρες στις οποίες δουλεύουμε. Και μια και δουλεύουμε εκεί, δεχόμαστε το γεγονός ότι φορολογούμαστε ε, επί των κερδών μας με ψηλότερους, πολύ ψηλότερους ε, φορολογικούς τελέσεις από ό,τι άλλες ε, βιομηχανίες. Δεν προσπαθούμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να μειώσουμε αυτούς τους συντελεστές. Ζητώ συγγνώμη. Όταν λέτε 53% κυρία μου, είναι ο εταιρικό φόρο αυτό μόνο, έτσι. Εκεί πάνω σε αυτό προστίθενται και άλλοι ειδικοί φόροι, ειδικοί για την παραγωγή. Όχι, μιλάω για τους, τη φορολογία επί των κερδών, έτσι. Ο φόρος της, πα, παραγωγής ε, είναι επιπλέον 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2014 μόνο, μας το είπατε αυτό. Ο 8,5 δισεκατομμύρια, 53% ε, συν 5 δισεκατομμύρια, που είναι εταιρικό φόρο, και το 5 δισεκατομμύρια που είναι επιπλέον φόρο. Φόρο παραγωγή. Τώρα, για τη διανομή. Το πώ κατανέμονται οι φόροι μα. Πολύ λογικά συνδέονται με τον τόπο που έχουμε τις δραστηριότητές μας και παράγουμε τα κέρδη μας. Γιατί η ευχή που ακούμε είναι ότι πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας εκεί που έχουμε τις δραστηριότητές μας. Έναν όμιλο όπως η Total Ακριβώς αυτό κάνουμε. Πολυλογικά, λοιπόν, το 55% των φόρων το πληρώνουμε στην Αφρική, γιατί έχουμε πολλές δραστηριότητε στην Αφρική, 20% περίπου στην Ευρώπη και το υπόλοιπο στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ευρώπη, κυρίως στην Νορβηγία πληρώνουμε τους φόρους, γιατί εκεί είναι η κυριότερη χώρα παραγωγός καθώς και στο Αμένο Βασίλειο και στην Ογκλανδία. Τώρα, να απαντήσω γιατί δεν πληρώσαμε φόρου ε, στα κέρδη που κάναμε στη Γαλλία το 12, 13 και 14. Γιατί, δυστυχώ δεν είχαμε καθόλου κέρδη. Είχαμε μάλιστα ζημίε. αρκετά σημαντικέ. Το 2011 πληρώσαμε επί των κερδών μας φόρους, γιατί είχαμε ε, κέρδη στη Γαλλία και δεδομένων των αποτελεσμάτων τον, το πρώτο τρίμηνο του 2015, θα πληρώσουμε μάλλον φόρους το 2015. Ο λόγος είναι απλός. Στη Γαλλία έχουμε δραστηριότητες κυρίως ε, δίληση, ε, πετροχημικές δραστηριότητε, ειδική χημεία. Αυτές οι δραστηριότητε όμω πλήττονται λόγω Ε, η τιμή του αργού πετρελαίου μέσα το 2012 επίσης έφτασε στα όρια ε, και ξεπεράσαμε τα, το περιθώριο κερδοφορίας ε, στη δίληση. Ε, πώς ανακάμψαμε, γιατί ανα, αναδιαρθρώσαμε τις δραστηριότητες δίλησης. Και επίσης ε, μειώθηκε πολύ η τιμή του αργού πετρελαίου και επομένως περισσότερα κέρδη ε, στα δηληστήρια. Επομένως ε, οι δραστηριότητες αυτές είναι πολύ ευαίσθητες στο, στη διακοιμάση των τιμών του αργού πετρελαίου και στην ισοτιμία με το δολάριο δεν έχει να κάνει με φορολογικές στρατηγικές, ας πούμε, επιθετικές κτλ. Έχει να κάνει με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο, στη δική μας, στο δικό μας κλάδο. Αυτό έτσι είναι μια, ένα πανόραμα για το πώς κατανέμονται οι φόροι μας. Άκουσα τις ερωτήσεις για τις θηγατρικές μας στην Ολλανδία και στους φορολογικούς παραδείσους. Να σας απαντήσω. γιατί λείπουν 30 θηγατρικές από τον κατάλογο που δημοσιεύσαμε. Δημοσιεύσαμε τον κατάλογο των θηγατρικών μας που είναι 903. Και καμιά τριανταριά θηγατρικές, δεν θυμάμαι ακριβώ, περίπου 30, που δεν αναφέρονται, είναι μη ενοποιημένες θηγατρικές, γιατί γιατί δεν είναι ουσιαστικέ σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητέ του, δεν έχουν καμία σημασία, είτε γιατί είναι οντότητε οι οποίε δεν έχουν πια ε, καμία δραστηριότητα και είναι σε φάση εκαθάριση, ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τη δραστηριότητά του. Επομένω, δεν είναι σημαντικέ για τον όμιλό μα. Γιατί ο κανόνα τη ενοποίηση ε, που χρησιμοποιούμε ε, και που τον ε, ελέγχουν οι λογιστέ μα είναι να μιλάμε για θηγατρικές που έχουν σημαντική επίπτωση, που είναι σημαντικές ε, στον όμιλό μας. Γι' αυτό ακριβώς δεν αναφέρονται 30 θηγατρικές. Γιατί τόσες ε, θηγατρικές στην Ολλανδία θα πρέπει να καταλάβετε τι δραστηριότητές μας γενικά. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε ε, μια δραστηριότητα εντάσσεως κεφαλαίου. πολύ συχνά χρειαζόμαστε να παρέμβουμε μαζί με εταίρου κτλ. Είναι κλασικό αυτό στον πετρελαϊκό τομέα. Ε, να δημιουργήσουμε δηλαδή μέσω άδειών μία οντότητα, ούτω ώστε και οι εταίροι μα να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ας πούμε, των δραστηριοτήτων μα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλέ διαφορετικέ νομικέ οντότητε, χωρί αυτό όμω να είναι αποτέλεσμα ε, προσπάθειας φορολογικής όπω όπως λέμε. Όχι, δεν γίνεται δεν εξοικονομούμε καν φόρους με αυτές τις πρακτικές εξάλλου. Και πολύ συχνά ε, έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει απλώς την εταιρική της έδρα Φερρυπίν στην Ολλανδία και όλη η δραστηριότητά της ε, γίνεται σε μια χώρα που παράγεται το πετρέλαιο ε, επειδή έχουμε πλατφόρμες πετρελαίου, επειδή έχουμε ε, εργοστάσια ας πούμε υγροποίησης κτλ. Ε, και πληρώνουμε εκεί φόρο γιατί εκεί έχουμε την, τις δραστηριότητε μας σε αυτές τις χώρες δηλαδή. Ε, γιατί έχουμε λοιπόν τώρα την εταιρική μας έδρα αλλού και κυρίως στη Γαλλία. Έχουμε διάφορες στην Ολλανδία βεβαίως, αλλά τις περισσότερες στη Γαλλία. Το Μάιο, ή μάλλον ε, βάζουμε την εταιρική έδρα σε μια χώρα όπως η Γαλλία ή η Ολλανδία. Γιατί? Γιατί πολύ συχνά στη χώρα όπου έχουμε τις δραστηριότητε μας πραγματικά, το δικαίωμα, το εταιρικό δίκαιο δεν μας επιτρέπει τέτοιου τύπου επενδύσεις. Ή αν δημιουργήσετε μία ε, εταιρεία τοπική, ας πούμε, βάσει το τοπικό δίκαιο, μας, μας υποχρεώνουν να την βάλουμε στο χρηματιστήριο στο, στο τοπικό νόμισμα και δεν έχουμε να την κεφαλαιοποιήσουμε στο τοπικό νόμισμα και δεν έχουμε αρκετό χρήμα, ας πούμε. Ε, δεν μπορούμε να, να φτιάξουμε λοιπόν ε, εταιρείε που να έχουν την έδρα τους εκεί γιατί κολλιόμαστε λόγω του, της κυκλοφορίας του χρήματος. Επομένως στη Γαλλία ας πούμε. Τώρα, γιατί το κάνουμε και στην Ολλανδία. Γιατί στην Ολλανδία μπορούμε να έχουμε ε, του, τα λογιστικά μας βιβλία σε δολάρια που είναι σημαντικό στην, στον τομέα μας, όπου κυρίως δουλεύουμε το δολάριο. Ε, να σας δώσω κάποια νούμερα τα οποία βρίσκονται και στα βιβλία μας. Συχνά αυτό το θέμα της, ε, των λογιστικών βιβλίων σε δολάριο ε, θεωρείται από τον κόσμο ως δικαιολογία. 10 ε, cent ε, αλλαγή της ισοτιμίας δολαρίου ευρώ έχει επίπτωση 1,65 δισεκατομμύρια στο, ε, στις δραστηριότητες, είχε μάλλον, στις δραστηριότητες Total το 2013. Είναι ε, τρομερό διακύβευμα αυτό. Ε, πρέπει να προστατευόμαστε όταν έχουμε αυτές τις α, τη α, της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ σχέση με το δολάριο και το να έχουμε τα λογιστικά μας βιβλία και τα φορολογικά μας βιβλία σε δολάριο είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος να προστατευτούμε απέναντι σε αυτές τις Άλλο παράδειγμα το οποίο έχω δώσει πολύ πρόσφατα στην γαλλική εφορία που με ρωτούσε για μια συγκεκριμένη εταιρεία μας στις Βερμούδες ε, διαπιστώθηκε ότι σε, ένα, σε μια θηγατρική που ε, είχαμε στις Βερμούδες η επίπτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αν είχαμε το, τα λογιστικά μας ε, σε ευρώ, θα ήταν πάνω από 100 ε, εκατομμύρια ευρώ. Ε, δεν το κάνουμε για φορολογική βελτιστοποίηση, αλλά γιατί έχουμε πρόβλημα πραγματικά λόγω φορολογικών διακυμάνσεων. λόγω Γιατί στην Ολλανδία λοιπόν, πριν πω στι Βερμούδε ή γενικά στου φορολογικού παραδείσου, πέρα από το γεγονό ότι αυτέ οι εταιρείε μπορούν να έχουν τα βιβλία του σε δολάριο, Πρέπει να γνωρίσουμε ότι στην Ολλανδία έχουμε σταθερή, σταθερό φορολογικό σύστημα, ένα νομικό πλαίσιο φορολογικό σταθερό, σημαντικό για τις δραστηριότητε μας. Επομένως, επιλέγουμε συχνά τις κάτω χώρες. Έχουμε αυτό το hub της χρηματοδότησης ε, ε, σε δολάριο και χρηματοδοτούμε ε, τις θηγατρικές μας παραγωγής πετρελαίου, α πούμε, που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Ε, τώρα, έχουμε λοιπόν την εταιρική μα έδρα στην ε, Ολλανδία. Όλα τα κέρδη βρίσκονται όμως, ε, παράγονται μάλλον στις χώρες που παράγουμε το πετρέλαιο και εκεί πληρώνουμε του φόρου. Ε, εάν πρέπει να σας πω μάλλον, ε, γίνεται μεγάλος λόγος για την εταιρική έδρα, αλλά φορολογικά δεν έχει καμία φορολογική επίπτωση. Ε, αν έχουμε απλώς την εταιρική μας έδρα σε μία χώρα, δεν γλιτώνουμε φόρους. Τώρα, άλλη ερώτηση. Γιατί έχουμε κάποιες εταιρείε στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι εταιρείε Αυτέ οι θηγατρικέ, οι 19 ας πούμε, για τις οποίες ε, σας αναφέραμε μέσω του καταλόγου μα δημιουργήθηκαν πριν από την ε, εξαφάνιση του γαλλικού φορολογικού καθεστώτος των επιημένων φορολογικών κερδών δηλαδή. Τα είχαμε δηλώσει δηλαδή στη γαλλική εφορία όλα αυτά, μπορεί να το επαληθεύσετε και η εφορία το επαλήθευσε, η γαλλική εφορία, και το αποτέλεσμα ήταν ότι συμπεριλήφθηκαν στα ε, φορολογικά στοιχεία της Total SA που φορολογείται στη Γαλλία. Δεν κάνουμε φορολογική βελτιστοποίηση ε, με το να βάλουμε ας πούμε ε, θηγατρικές στην Παχάμες Φελπίν. Σημαντικό να το υπενθυμίσω. Υπάρχει ευελιξία. Είχαμε απλώς λογιστικά βιβλία σε δολάρια, είχαμε ένα εταιρικό δίκαιο ευέλικτο στις Βερμούδες, μερικές φορές μπορεί να αγοράσει ένα νόμιλο εταιριών, συνολικά. Χρειάστηκε, το έχουμε κάνει δηλαδή. Και ο προηγούμενος αγοραστής είχε ε, επιλέξει να είναι κατευθυμένος στι Βερμούδες, για δικούς του λόγους. Όχι για λόγους δικού μα της Total, αλλά δεν είναι και εύκολο να επαναπατρίσουμε την εταιρική έδρα και να αλλάξουμε έτσι από ενία νυχτή Έχουμε μία πλειάδα λοιπόν λόγων για τους οποίους ε, μπορούμε να βρισκόμαστε στις Βερμούδες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο στόχος μας είναι να κάνουμε φορολογική βελτιστοποίηση. Δεν ξέρω ποια ήταν τα υπόλοιπα ερωτήματα. Τώρα, για το θέμα των φορολογικών παραδείσων και γιατί λέμε ότι έχουμε μόνο 19 εταιρείε ενώ Ορισμένοι κατάλογοι φορολογικών ε, παραδείσων ε, συμπεριλαμβάνουν 80 χώρες και το καθεξής. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι κάποιοι είχαν την αξιοπιστία τους ε, καταρτίζοντας καταλόγους όπως είναι και στο Tax Justice Network 80 χώρες όπου έχουμε και Γερμανία, Βέλγιο και το καθεξής. Νομίζω ότι πολλοί δεν αξιοποιούν αυτό τον κατάλογο των 82 χωρών, αλλά παλαιότερο, πολύ πιο περιορισμένο κατάλογο, το οποίο πλήρει περισσότερο τα κριτήρια, τα γενικά, για το τι θεωρείται προλογικό παράδεισο. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το γεγονό ότι δεν υπάρχει συνένεση επενό του καταλόγου φορολογικών παραδείσων. Και εμεί χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα κατάλογο, παρότι έχει και αδυναμίες. Θα μπορούσε να βελτιωθεί. Όμως ε, αυτή η έλλειψη καταλόγου δημιουργεί πρόβλημα. Γι' αυτό και η Total επέλεξε να δημοσιεύσει το κατάλογο το θεατρικό της, γιατί έτσι μπορεί ο καθένας με βάση τη δική του αντίληψη του τι συνιστά φορολογικό παράδεισο να ε, τα εξετάσει όλα αυτά τα στοιχεία. Εμείς έχουμε 19 ε, εταιρείε στις χώρες που συνήθως θεωρούνται ως φορολογική παράδειση. Όσοι θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλοι φορολογική παράδειση, βεβαίως μπορούν να σχηματίσουν την άποψή τους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αν θεωρούν ότι πρέπει να επικρίνουμε και άλλες χώρες, ε, έχουν το δικαίωμα να το θίξουν. Πολύ σημαντικό ζήτημα, όπως ανέφερε και ο συνάδελφός μου την Παριμπά, είναι το θέμα της επίλυσης διαφορών. Και εδώ είναι κάτι που μας προβληματίζει. Αύξηση των περιπτώσεων διπλής και πολλαπλής φορολόγησης. Θεωρούμε ότι οι εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο του BEPS ε μπορούν αναπόφευκτα να οδηγήσουν στην, στον παραπλησιασμό αυτών των διαδικασιών. Γιατί έχουμε τις ε, γενικές διεθνείς ε, αρχές φορολόγησης, χωρίς όμως να έχουμε και μία συνένεση μεταξύ των χωρών για το ποιοι θα είναι μελλοντικοί κανόνες και ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει συνένεση σε ό,τι αφορά την, και τη δέσμευση των ε, χωρών να εφαρμόσουν ε, τους κανόνες BEPS. Επομένω, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν διαφορετικέ ερμηνείε, στρεβλώσει στην εφαρμογή από τη μία την άλλη χώρα και έτσι θα έχουμε πολλαπλασιασμό ε, των περιπτώσεων πολλαπλή φορολόγηση. Αυτό είναι κάτι που μα ανησυχεί ιδιαίτερω, γιατί ο μηχανισμό ε, εξάλληψη αυτή τη διπλή φορολόγηση αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σωστά. Δεν είναι αποτελεσματικό. Και θεωρούμε ότι τα, οι χώρε που θα υιοθετήσουν τον BEPS θα έπρεπε τουλάχιστον να δεσμεύονται εν είδη αντισταθμίσματος να ε, εξαλείψουν ε, αυτή την διπλή φορολόγηση και να δεχθούν να μειώσουν τη δική τους φορολογική βάση σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι δύο ακόμα σε μία μένουν για το CCCB. Για το πρώτο λοιπόν, την ε, κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση εμείς θεωρούμε ότι η ενοποίηση που κάναμε παγκοσμίω ήταν ένα πολύ καλό μέσο καταπολέμησης ε, της ε, μεταβίβασης φορολογικής βάσης από τη μια χώρα στην άλλη. Βεβαίως ε, ήταν καλό να γίνει αυτή και στις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως βεβαίως έτσι θα αποτρέψουμε και τις μεταβιβάσεις εκτός Ένωσης για τις ε, εκθέσεις αναχώρα τώρα. Εμείς βεβαίω δεν είμαστε αντίθετοι με τη διαφάνεια. Από μόνοι μας δημοσιεύσαμε τον κατάλογο των θεατρικών μας. Επίσης έχουμε κοινοποιήσει στη Γαλλική Φορολογική Αρχή όλα τα στοιχεία που αφορούν τις θεατρικέ μας ανά τον κόσμο, για να μην υπάρχει δηλαδή δεν μα προβληματίζει δηλαδή το να θέσουμε επιτάπητο αυτά τα στοιχεία και να τα δώσουμε και στις φορολογικές αρχέ, όμω από την άλλη τι μα προβληματίζει Επανέρχομαι σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Ε, μία ανεξέλεγκτη τέτοια μεταβίβαση στοιχείων ε, και ε, το ενδεχόμενο θέμα του ανταγωνισμού ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ότι δηλαδή κάποιοι θα πρέπει να τηρούν αυτή την υποχρέωση για το κριτήριο, ενώ άλλοι όχι. Εκεί λοιπόν υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού και όταν αυτά δημοσιεύονται, βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα να δημοσιεύονται και να γίνεται και κατάχρηση. Σας ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποια ερωτήματα να θέσω και βλέπω ότι και ο εισηγητής ε, θέλει να πάρει το λόγο στη συνέχεια. Για το τελευταίο αυτό σημείο, αν κατάλαβα καλά, υπάρχει μία διαφορά διάσταση απόψεων σε ό,τι αφορά τις εκθέσει αναχώρα, γιατί από πλευρά τραπεζικού τομέα όλα δημοσιοποιούνται. Και δεν διαπιστώθηκε ότι αυτό στρεβλώνει τόσο τρομερά τον ανταγωνισμό σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ναι, αν με επιτρέπετε, ίσως να μην αναφερόμαστε στην ίδια διαδικασία υποβολής εκθέσεων αναχώρα, γιατί το περιεχόμενο ε, ε, των εκθέσεων αναχώρα στις τράπεζες δεν είναι το ίδιο. Ήταν πολύ πιο περιορισμένο σε σχέση με τον BEPS. Δηλαδή, μια υποβολή εκθέσεων αναχώρα με βάση το μοντέλο που ισχύει στις τράπεζες, ε, δεν θα μας ανησυχούσαμε, δεν μας προβλημάτιζε. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι. Αυτό το σημείο. Ε, το κύριο, τα κύρια στοιχεία που έχουμε στα τραπεζικά πρότυπα είναι κάτι το οποίο επανέρχεται και στο πλαίσιο του ΩΣΑ. Βεβαίως, δεν δημιούργησε σημαντικά προβλήματα. Τώρα η κατάσταση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας. Είναι δύσκολο να το αξιολογήσει κανείς. Όμως θεωρώ ότι τα δύο πρότυπα και από πλευράς ΟΣΑ και στον τραπεζικό τομέα δεν διαφέρουν και τόσο πολύ. Ωραία, ευχαριστώ. Κάτι ακόμα για τις Βερμούδες. Αν κατάλαβα καλά. Για ιστορικούς μάλλον λόγους έχετε θηγατρικές εκεί. Αναφέρομαι στις Βερμούδες γιατί μάλιστα και αύριο θα έχουμε ε, και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό των Βερμούδων που θα έρθει εδώ. Γι' αυτό θα ήθελα να προετοιμαστώ και εγώ να έχω πιο συγκεκριμένα ερωτήματα να του θέσω. Για ιστορικού λόγου λοιπόν, γιατί υπήρχε και προηγούμενη εταιρεία ε, που Είχε την έδρα εκεί και στην περίοδο που το γαλλικό σύστημα προβλέπει αυτή την ενοποιημένη φορολογική βάση δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα διαφάνειας γιατί είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι δραστηριότητές σας ε, όμως αυτό δεν ισχύει σήμερα. Παραμένετε όμως στους Βερμούδες για αυτούς τους ιστορικούς λόγους και στις Βερμούδες και άλλου. Ναι, να σας απαντήσω. Πράγματι για ιστορικούς λόγους μάλιστα σε ορισμένε περιπτώσει ε, αυτοί οι λόγοι ανάγονται στη δεκαετία του 50. γιατί τότε δεν ήταν ε, σκόπιμο μία γαλλική εταιρεία να ε, εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνει τις αστριότητες της σε δολάρια. Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, έχουμε και συγκεκριμένο άρθρο του Γενικού Φορολογικού Κώδικα, δηλαδή αν, υπάρχει, αν υπάρχουν ευνοϊκέ διατάξεις, ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο που μας οδηγεί να πληρώνουμε λιγότερο από το ίμιση των φόρων ε, στις Βερμούδες, Βεβαίω όλα αυτά τα δηλώνουμε και εξακολουθούμε να τα δηλώνουμε και στις γαλλικές φορολογικέ αρχές. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι αυτό εύκολα και πολύ αποτελεσματικά ε, διασταυρώνεται. Μετά θέλαμε να αποσύρουμε όλες ε, τις, ε, να αφαιρέσουμε από την επικράτεια των Ευρωμούδων όλες τις εταιρείες που μπορούσαμε. Μας έμειναν ε, περίπου 10 γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν. Επειδή είχαμε μόνο 13% για παράδειγμα συμμετοχή στις, ε, μετοχή, στις εταιρείες αυτές σε αυτές τις περιπτώσεις ε, μπορεί να γίνει μόνο μέσω ε, ρευστοποίησης ή παραχώρησης. Εκεί λοιπόν θεωρούμε ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία φοροδιαφυγή στις Βερμούδες και όλα αυτά δημοσιεύονται και κοινοποιούνται στις γαλλικές αρχές, δεν ε, αξίζει τον κόπο να μπούμε σε αυτό το ρίσκο και να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. 14 είχαν ε, μεταφερθεί στο τέλος του 2014 και ακόμα 3 μέχρι τα τέλη του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ που ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μας για να κατανοήσουμε και εμείς πώς ακριβώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί της απορρόφησης, ε, της συμμετοχής σε κάποιες εταιρείες που ε, έχουν την έδρα τους σε μια επικράτεια και έχουν και δικαίωμα εξόριξης σε ορισμένες περιπτώσεις. δεν μιλώ για άλλες κατηγορίες όπως ε, πνευματικών δικαιωμάτων και το καθεξής. Αναφερθήκατε στην περίπτωση της Ολλανδίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε αυτό το ερώτημα την επόμενη εβδομάδα με ένα δεύτερο πάνελ στην Airbus. Η Έστρεντε Λάγκε και άλλοι Ολλανδοί συνάδελφοι παρευρίσκονται. Εγώ νομίζω και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ότι έχουμε εκεί πολύ συγκεκριμένο εταιρικό δίκαιο που επιτρέπει σε συγκεκριμένε επιχειρήσει να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξία σε σχέση με άλλε νομιστικέ διατάξει. Και έτσι, αν μια επιχείρηση αποφασίσει και επιλέξει να θέσει την έδρα τη σε μία χώρα αντί άλλη, μπορεί να υπάρχουν και φορολογικέ προεκτάσει. Και όπω ίσω αναφέρατε και στο πλαίσιο τη δική σα δραστηριότητα, το γεγονό ότι κάποιο έχει κοινωνική εταιρική έδρα σε μία ε, χώρα δεν έχει καμία φορολογική επίπτωση. Αυτό δεν αφορά τη δραστηριότητα. Όμως στην Ολλανδική περίπτωση θα ήταν καλό να το διαρευνήσουμε αυτό και πιο συγκεκριμένα με την Airbus. Κύριε Τόιρερ, θέλετε να επανέλθετε, να δευτερολογήσετε. Η κυρία, ε, ε, όπως απάντησε για την πολιτική της Total για την ε, υποβολή εκθέσεων. Μα απάντησε, λέει ο πρόεδρος. Με συγχωρείτε, λέει εκπρόσωπος της Total. Εγώ νόμιζα ότι απάντησε, αλλά κάτι δεν άκουσα. Χωρίς μικρόφωνο, η κυρία Γκόμες επαναλαμβάνει την πολιτική της Total για τι ε, εκθέσεων από Μα Το είπε λέει η πρόεδρος. Η εκπρόσωπο της Total. Δεν ε, αντιτιθέμεθα στην υποβολή εκθέσεων χώρα. Αλλά, όχι, να το πω αλλιώ, μέσω αυτών των εκθέσεων για τα ενοποιημένα κέρδη δίνουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στις γαλλικές φορολογικές αρχές. Αλλά λοιπόν αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι απαιτείται πολύ αναλυτική παρουσίαση στοιχείων στα πρότυπα που προτείνει το BEPS και επίσης στρέβλος ανταγωνισμού που θα μπορούσε να προκύψει εάν μόνο κάποιες χώρες, μόνο κάποιες επιχειρήσεις έχουν αυτή την υποχρέωση. Να σας πω λοιπόν κάτι παραπάνω γιατί κάποιες πληροφορίες μπορεί να είναι ευαίσθητες. Για παράδειγμα, αν έχετε 25 θηγατρικές σε μια χώρα με διαφορετικές δραστηριότητες η ενοποίηση αναχώρα δεν θα επιτρέψει στους ανταγωνιστές σας να ε, μάθουν εμπιστευτικά στοιχεία. Αλλά αν είναι πολύ ανταγωνιστική κατάσταση με για παράδειγμα διαγωνισμούς όπου έχετε μόνο μία θηγατρική σε μια χώρα η ε, δημοσίευση πληροφοριών για αυτή τη μία θηγατρική θα δώσει ανταγωνιστές σας πληροφορίες για τις δομές σας, ε, τη λειτουργία σας, την πολιτική τιμών σας. Για παράδειγμα, ε, επιχειρήσεις που έχουμε στην ίδρυυση φοβούνται ότι αυτό μπορεί να δώσει πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση σε άλλες εταιρείε για την πολιτική τιμών τους, και για το πώ προτίθενται, για παράδειγμα, να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό για δημόσιες προμήθειε, Φοβούνται λοιπόν, για παράδειγμα, ότι μπορεί να προτείνει να μειοδοτήσει κάποιο ανταγωνιστής του. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος, Τόιρερ και μετά ο κύριο Μαραγάλ για του πράσινου. Τόιρερ. Πρέπει να ομολογήσω ότι η απάντησή σα για την παρουσία σα στι βερμούδε δεν ναι, με έπεισε, ξέρετε. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Αλλά δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο νησί της Καραβικής όπου έχετε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Υπάρχει πολύ καλή... Ε, υπάρχει ε, πολύ παλό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. Μάλλον πιο πιθανό ότι έχει πολύ ωραίες παραλίες. Για ποιο λόγο χρειάζεται να είστε παρόντες εκεί. Είπατε ότι είναι παλιά παράδοση κάποτε που δεν υπήρχαν ανοιχτέ αγορέ. Αλλά ξέρετε αυτές είναι επικράτειες όπου είναι πολύ καλές συνθήκες για υπεράκτιες δραστηριότητε. Διότι κατά τα άλλα οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για να καταστήσεις μια επιχείρηση. Μόνο αν θέλεις να υποφεληθεί από κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις από πλευράς φορολογίας, από πλευράς ελέγχου των δραστηριοτήτων σας, η εκπρόσωπος... Α, όχι, κυρία Φερέιρα. Ναι, επ' αυτού ακριβώς. Νομίζω ότι κατάλαβα εν μέρη τη λογική σας αλλά δεν θα έπρεπε κάπως να διευκρινίσετε και εσείς και η Παριμπά τη στρατηγική σας σε σχέση με αυτές τις δικαιοδοσίες. Αν θέλετε να φαίνεστε και θα έπρεπε να θέλετε να φαίνεστε ότι συμμορφούστε τότε εάν δεν δώσετε καλές εξηγήσεις για την παρουσία σας σε αυτές τις ε, περιοχές Αφισβητείτε η συνολική σα στρατηγική. Είναι κακό για την υπόλοιψή σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα διαφανείς στις εξηγήσει σα. Πρέπει να επιμείνουμε πιστεύω λοιπόν. Πρόεδρος, περιμένετε, περιμένετε κυρία μου. Να πάρουμε και την του κυρίου Μαραγάου από τους Πρασίνους που δεν μπόρεσε να εκφραστεί. Δεν ήταν εδώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με συγχωρείτε γιατί δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα. Συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ελπίζω τώρα να μην επαναλαμβάνω ήδη υποθέντα. Πρώτον, για το θέμα των θηγατρικών στην Ολλανδία. Άκουσα τις τελευταίες εξηγήσεις για τις 30 που δεν αναφέρονταν στο κατάλογο. Εκτός από αυτές, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις αυτή η δομή με θυγατρικές θυγατρικών που δεν αφορά μόνο την χώρα όπου έχουν την εταιρική τους έδρα αλλά τη δραστηριότητα σε άλλες χώρες για παράδειγμα στην Ουγκάντα σε μια περίπτωση στην Ιγυρία υπάρχει μια σαφής τέσσερα επίπεδα θυγατρικών η μία της άλλης που, καθ, που συνδέουν τη δραστηριότητα της Total στην Ολλανδία με τη δραστηριότητά της στην Ιγυρία. Πώς το εξηγείτε αυτό. Δεύτερον, υπόθηκε αλλά θέλω να επιμείνω. Η Total γιατί δεν στηρίζει πλέον αυτή την πρόταση για μια ενοποιημένη βάση εταιρικού φόρου. Διότι μέχρι πρόσφατα, πρόσφατα τη στήριζε. Πρόσφατα ο πρόεδρος ανήγγειλε αυτή την αλλαγή στάσης. Για παράδειγμα, τι φόρους πληρώνετε στη Γαλλία, που είναι η φυσική σα α πούμε μέτρα. Το 12, 13 και 14 δεν πληρώσατε στη Γαλλία φόρους. Παρά το ότι είχατε κέρδη που δηλώσατε τι εταιρείε του ομίλου 15,8 δι δολάρια το 12 και 14,3 το 13. Η επίσημη εξήγηση είναι ότι δεν υπήρχαν κέρδη στην ε, Γαλλία. αλλά ο πρόεδρος ε, Πατρίκ Μπουγενέ είπε ότι ε, από τούτο και στο εξή θα πληρώνει στη Γαλλία φόρο από το 2015 και μετά. Τι άλλαξε από τη μια χρονιά στην άλλη. Γιατί άλλαξε έτσι η στάση σας. Γιατί δεν είδα καμία ουσιώδη αλλαγή στην κερδοφορία σας. Γιατί προηγουμένως δεν ήταν κέρδη και τώρα ξαφνικά είναι. Μήπως έχει να κάνει αυτό με θέματα φοροδιαφυγής. Και τέλος, θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα. Για την αντίθεσή σας στην υποβολή εκθέσεων αναχώρα, για λόγους ανταγωνιστικότητας. Επειδή να μειώσετε την ανταγωνιστικότητά σα ε, έναντι άλλων εταιριών που δεν θα υποβάλλουν τις εκθέσει. Θα ήθελα περισσότερη σαφήνεια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Ορισμένε ερωτήσει έχουν ήδη απαντηθεί, αλλά θα μπορούσατε να επανέλθετε γρήγορα. Τελευταίο ο μιλητή ο κύριο Ντεμαζή. Φάμπιο Ντεμαζή. Τομάση, συγγνώμη διευκρίνηση θα ήθελα. Ο εκπρόσωπος της Total δεν απάντησε για το τι ποσοστό των κερδών περνάει από την Ολλανδία. Και δεύτερον, σας κατάλαβα καλά, κύριε εκπρόσωπε της BNP ε, Paribas, είπατε ότι κατά τη γνώμη σας οι εκθέσεις αναχώρα που θα ήταν υποχρεωμένη η Total να ακολουθήσει σύμφωνα με την BEPS και που είναι παρόμοια με αυτά που κάνουν οι τράπεζες. Και τώρα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Total, σε πόσα από τα 28 κράτη-μέλη θα είχατε δυνατότητα να έχετε λογαριασμούς ε, σε δολάρια. Ευχαριστώ που μπορώ να επανέλθω για το θέμα των Βερμούδων, γιατί έγιναν τόσες ερωτήσεις που Ίσως ε, δεν ήμουν επαρκώς λεπτομέρης. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τόιρα. Οι Βερμούδες δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένες υποδομές. Αλλά η θέση μας είναι απόλυτα συνεπής. Στις Βερμούδες έχουμε μόνο την εταιρική έδρα ενός νομικού προσώπου δικαίου. Και δεν προκύπτουν κέρδη από τη δραστηριότητά μας στις Βερμούδες. Το πρόβλημα μπορεί να είναι ε, να μεταφέρονται κέρδη στις Βερμούδες όπου δεν υπάρχει δραστηριότητα. Εμείς δεν έχουμε κέρδη στις Βερμούδες. Γιατί όμως έχουμε εταιρείες. Γιατί στο παρελθόν υπήρχε αυτό. Ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχαν έλεγχοι στην ε, κυκλοφορία των κεφαλαίων. Γι' αυτό είχαμε εκεί εταιρείε που μπορούσαν να λειτουργήσουν σε δολάρια. Και επίση επειδή είχαμε αγοράσει εταιρείε που ήταν, είχαν εδώ Τώρα, για το ενοποιημένο κέρδο μα στη Γαλλία, αφαρμόσαμε του ίδιου κανόνε από το 1966 με το 2010. Όλε μα οι εταιρείε δηλώνονταν και φορολογούνταν στη Γαλλία. Δηλώνονταν στι γαλλικέ φορολογικέ αρχέ. Δεν είχαμε κανένα φορολογικό πλεονέκτημα έχοντα την ε, εταιρική μα έδρα εκεί. Μέχρι το σημείο θα μπορούσα να πω που. Εντάξει, τώρα συνοψίζω. Η Total δεν είχε κανένα συμφέρον. Θα μπορούσαμε να αγνοούμε ότι είναι φορολογικό παράδεισο. Πληρώναμε φόρου στη Γαλλία. Πολλέ φορέ χρειάστηκε οι γαλλικές φορολογικές αρχές να δώσουν πιστοποιητικά έναντι άλλων φορολογικών αρχών που ανησυχούσαν για αυτές μας τις έδρες για να επιβεβαιώσει ότι όλα μας τα κέρδη δηλώνονταν στη Γαλλία και περιέχονταν στην ε, φορολογητέα μας βάση. Είχαμε νομικά πλεονεκτήματα μέσω των εδρών μας στις Βερμούδες, αλλά δεν είχαμε φορολογικά πλεονεκτήματα. Αυτή ήταν το παρελθόν. Αυτή ήταν η κατάσταση στο παρελθόν, όπως είπε ο κύριος Λαμασούρ. Τώρα αυτά τα ενοποιημένα κέρδη καταργήθηκαν. Δηλαδή η διάταξη για τα ε, ενοποιημένα κέρδη. Γι' αυτό θέλουμε τώρα να καταργήσουμε τις εταιρείες μας τις Βερμούδες γιατί θέτουν προβλήματα υπόλοιψη παρά το ότι δεν κερδίζουμε τίποτα. Η λογαριασμοί, οι τραπεζικοί λογαριασμοί αυτών των εταιριών δεν είναι στις Βερμούδες, ε, τις περισσότερες φορές είναι στη Γαλλία. Και βεβαίως οι αρχές, ε, οι ελεκτικές για τα λογιστικά μας μας δίνουν τις αναγκαίες πιστοποίησεις. Στο παρελθόν είχαμε κατασταθεί για άλλους λόγους, όχι φορολογικούς. Δεν είχαμε κέρδη εκεί. Σήμερα επειδή δημιουργεί ερωτηματικά για θέματα υπόλοιψης, το καταλαβαίνουμε, ανταποκρινόμεθα λοιπόν σε αυτήν την απέτηση κοινή γνώμη και επαναπατρίζουμε τι περισσότερε εταιρείε από αυτέ τι χώρε. Και δεν ανοίγουμε καινούριε, πρόεδρο. Δηλαδή θα καταργήσετε ή θα επαναπατρίσετε όλε όσε έχετε στι Βερμούδε. Ναι, ναι, ναι, ναι, είμαστε στην πορεία. Είμαστε στην πορεία. Από το 12, 14, 14 νομικά πρόσωπα έχουν ε, επαναπατριστεί στην Γαλλία ή άλλε ευρωπαϊκέ χώρε οι περισσότερες στη Γαλλία, οι πολύ περισσότερες. Τρεις ακόμη είναι σε φάση ε, μεταφοράς. Μέχρι τις 30 Ιουνίου ελπίζουμε να εγγραφούν στα Μητρώα τα αντίστοιχα και ελπίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου να λήξουν και οι υπόλοιπε έξι, δηλαδή να λήξει η παρουσία τους εκεί. Θα μείνουν 9-10 για τους οποίες από νομική πλευρά δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε αυτόν τον επαναπατρισμό. Για τα άλλα σημεία. Άκουσα το ερώτημα για τις σχέση διοκτησίας της εταιρείας που έχουμε στην ε, Νιγηρία, ότι υπήρχαν τέσσερα επίπεδα στην Νιγηρία, στις εταιρείες αυτές. Ε, ο αριθμός των ενδιάμεσων ε, θυγατρικών δεν οδηγεί σε φοροδιαφυγή η Total έχει προκύψει ε, από συγχώνευση μεταξύ Total και της ΕΦ. Υπάρχει μία νομική οντότητα που είναι η ΑΛΦΑ Κιτέν. Για λειτουργικούς λόγους αποφασίσαμε να διαρθώσουμε τα διάφορα, ε, τις διάφορες μας σε holding γαλλικού τύπου. Έχουμε τρεις γαλλικές εταιρείες ε, ε, αμυγός γαλλικές ανάμεσα στην Τοτάλεσσα και σε όλες τις θηγατρικές μας, είναι τα ενδιάμεσα επίπεδα, και έχουμε στην Ιγυρία ε, διάφορες εταιρείε ε, νιγηριανού δικαίου. Μπορεί να υπάρχει και μια γαλλική, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Μπορώ να το επαληθέσω και να σας δώσω την απάντηση. Δεν γίνεται καμία φορολογική πάντως βελτιστοποίηση ε, λόγω του γεγονός ότι έχουμε αυτή τη διάρθρωση ε, μεταξύ της ε, Total SA που είναι η επικεφαλής της εταιρείας μας και των δραστηριοτήτων μας στην Νιγηρία ή στην Καμπών. Δεν κατάλαβα το ερώτημα για το ότι η Total δεν υποστηρίζει πια το project ενιαίας φορολογικής βάσης. Το υποστηρίζαμε και μετά είπαμε ότι είμαστε κατά. Η Total μάλιστα θα συμμορφωθεί και είναι υπέρ των προσπαθειών αυτών συντονισμού και εναρμόνισης που γίνονται στο εσωτερικό της Ένωσης και μάλιστα και εκτός αυτής. Δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι στο να υπάρχει μια κοινή φορολογική βάση και στις ειδικέ αναχώρα εκθέσεις. Είπαμε ότι προφανώς αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση θα συμμορφωθούμε. Και ξέρω στον εξωτερικό κλάδο υπήρχε μια τέτοια υποχρέωση στη Γαλλία. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα υπάρχει και για την οικονομική χρήση του 2015 και είμαστε έτοιμοι να συμμορφωθούμε. Λυπόμαστε όμως που μόνο οι γαλλικές εταιρείε και οι βρετανικέ εταιρείε έχουν αυτή την υποχρέωση και σήμερα οι Αμερικάνοι συνάδελφοί μα, α πούμε ε, δεν υφίστανται κάτι τέτοιο. ο νόμος Dodd-Frank, ο οποίος είχε ξεκινήσει να, και ήθελε να του επιβάλλει κάτι τέτοιο, έχει ανασταλεί. Εμείς πάντως θα συμμορφωθούμε. Για τον εταιρικό φόρο στη Γαλλία απάντησα. Ο κ. Μαραγκάλ έδωσε μια, έθεσε μια ερώτηση ότι επί πολλά χρόνια δεν πλήρωσε το τάλ φόρο στη Γαλλία. Κύριε Μαραγκάλ, η κυρία Μονιετή σας εξήγησε ότι η δραστηριότητα της Total στη Γαλλία είναι η δίληση. Η δραστηριότητα στη Γαλλία ήταν ελληματική όταν είχαμε, αλλάξαν οι τιμές ας πούμε, στο βαρέλι. Γι' αυτό δεν πλήρωσε εκείνες τις χρονιές. Νομίζω, δηλαδή δεν είχε κέρδη εκείνες τις χρονιές. Λοιπόν, απάντησαν οι εταιρείε. Ε, μας δώσατε και γραπτά σχόλια, μας απαντήσατε και προφορικά με πολλές λεπτομέρειες σε όλες τις ερωτήσεις των ε, Ευρωβουλευτών. Σας ευχαριστώ. Θα σας ε, απελευθερώσω. Η συνεδρίαση μας βέβαια είναι δημόσια και αν θέλετε μπορείτε να παραμένετε στην αίθουσα. Σας προτείνω τώρα να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης που είναι ο απολογισμός από τις έρευνές μας και από τις έξι αποστολές που κάναμε επιτόπου την περασμένη εβδομάδα, 18 Ιουνίου, μέσω, επισκέψη, μέσω μιας επίσκεψης στο Λονδίνο. Νομίζω ότι είναι καλό και το ήθελαν και οι συγητές να δούμε πώς πήγανε τα πράγματα. Το πρώτο τμήμα των εργασιών μας, δηλαδή, που ήταν να συλλέξουμε διάφορες, διάφορο, διάφορες πληροφορίες, ε, τεκμηρίωση, υλικό κτλ. μέσω των ακροάσεων, έτσι, όπως τη σημερινή ας πούμε, και έχουμε οργανώσει πολλοί άριθμες τέτοιες ακροάσεις. Έχουμε και μία σειρά ακροάσεων την επόμενη εβδομάδα 2 Ιουλίου, μια σημαντική χρονική στιγμή για μας, γιατί θα ξεκινήσουμε τη μέρα με μια μεικτή συνεδρίαση της δικής μας ε, Επιτροπής με την Οικονομική Επιτροπή για να γίνει μια ακρόαση με τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ και τον επίτροπο Μοσκοβισή που θα μας παρουσιάσουν το πακέτο του σχεδίου δράσης που υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εν συνεχεία θα έχουμε το πάνελ με τους ομιλητές ε, με ομιλητέ από τις, τον κόσμο των επιχειρήσεων και θα είναι παρούσα και η Airbus. Λάβαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό απαντήσεων στο ερώτημα στο ερωτηματολόγιο που στείλαμε στους 28 υπουργου Οικονομικών. Είμαστε σε φάση εξέτασης των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο. Λάβαμε επίσης απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λάβαμε απαντήσεις γραπτές, συμπληρωματικέ από τους μεγάλους τέσσερις και από άλλες προσωπικότητες ε, που ρωτήθηκαν εδώ, είτε εδώ στην Επιτροπή Τάξ, είτε στις ε, επισκέψεις που κάναμε τόπου. σε ό,τι αφορά τους υπουργούς, είμαστε σε μόνιμη επαφή και διαπραγμάτευση για να λάβουμε κάτι που δεν έχουμε λάβει ακόμα, πηγαίνοντας να τους δούμε. Να έρθουν δηλαδή τι, δεν έχουμε πετύχει, να έρθουν εδώ ενώπιον τη επιτροπή μα για να παρουσιάσουν τη θέση του οι υπουργοί αυτοί. Την κατάσταση τη χώρα του σε ό,τι αφορά την φορολόγηση των επιχειρήσεων και τη θέση τους ό,τι αφορά το πακέτο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη θέση του επί του σχεδίου δράση του ΟΣΑ. Δεν μπορώ να σα πω περισσότερα τώρα, γιατί είμαστε σε φάση διαπραγμάτευση ακόμα με τους υπουργού, αλλά είμαι αρκετά αισιόδοξο ότι υπάρχει δυνατότητα να συγκατατεθούν και να έρθουν 38 ονόματα εδώ που θα μας επιτρέψουν να ακούσουμε απόψεις πολύ διαφορετικές για να έχουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Μάλιστα, μετά από αυτά, καλό θα ήταν να δούμε τι πρώτες εντυπώσεις συλλέξαμε και τι διδάγματα από τις πληροφορίες που έχουμε λάβει μέχρι τούδε, από τις ε, επιτόπιες επισκέψεις μας. Επισκεφθήκαμε έξι χώρες, το Βέλγιο πρώτο, Λουξεμβούργο μετά, Ιρλανδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλες τις περιπτώσεις, σε κάθε περίπτωση, οι επισκέψεις αυτές ε, διεξήχθησαν όπως ακριβώς είχαν προβλεφθεί. Ευχαριστώ τη Γραμματεία γιατί στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπήρξε τέτοιο παράδειγμα επιτροπής μόνιμης ή προσωρινής που κατάφερε να στείλει, να κάνει έξι αποστολές, έξι επισκέψεις δηλαδή, σε έξι εβδομάδες σε διαφορετικές χώρες. Κάθε φορά λοιπόν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής υπουργό, με την φορολογική αρχή, τις φορολογικές αρχές, τους ε, εκπροσώπους της Βουλής που παρακολουθούν τις, τα φορολογικά θέματα, τους εκπροσώπους του τύπου, των καταγγελόντων, των whistleblowers, του επιχειρηματικού κλάδου, των μεγάλων γραφείων ορκωτών λογιστών, ακαδημαϊκούς και άλλους που μας επέτρεψε να πάρουμε πραγματικά μια πολύ καλή ιδέα για το τι συμβαίνει στις χώρες αυτές. Οι συντονιστές θα ήθελα να ξεκινήσουν πρώτοι να μας πούν και είναι εντύπωση που αποκόμισαν. Καταρχάς εννοώ την Ελίζα, βέβαια την εισηγήτρια. Ναι, μπορώ να επιβεβαιώσω τα όσα είπατε. Τώρα έχουμε μία, ένα σημαντικό όγκο διαθέσιμων πληροφοριών. Ουσιαστικά θέλαμε να καλύψουμε πολιτικές οντότητες, αξιωματούχους του φορολογικού συστήματος, εμπειρογνώμονες, μη κυβερνητικές οργανώσεις συμβούλους και ακαδημαϊκούς ερευνητές. Σε αρκετές περιπτώσεις ε, επισκεφθήκαμε και το Κοινοβούλιο και κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σε σχέση με αυτές τις πολιτικές οντότητες και Είδαμε και πώ ακριβώ δεξάγεται αυτή η συζήτηση στο ιστορικό κάθε κράτου μέλους και τη Ελβετία, βέβαια. Μα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη σαφώς και βλέπουν ε, τα θέλγητρα των άμεσων ξένων επενδύσεων και γενικά επιχειρηματικής δραστηριοποίηση και φορολογητέου εισόδηματο ως βασικού, κανόνας, βασικού κανόνα. Και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών για να είναι ελκυστικές και να προσελκύσουν δηλαδή <coughs> τέτοιες ε, εταιρείε για να έχουν φορολογητό εισόδημα. Βλέπουμε ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω τι ε, φορολογικέ συμφωνίες. Αυτά τα rulings έχουν ένα διτό χαρακτήρα. Αφενό έχουμε το σύνηθες επιχείρημα ότι απλώς επιβεβαιώνουν τους νόμους ότι οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν να αλλάξουν τους νόμους, απλώς τους επιβεβαιώνουν λοιπόν. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, των επιχειρήσεων, παρέχει και περαιτέρω σταθερότητα. Θεωρείται λοιπόν μια καλή ε, πρακτική συνεργασία μεταξύ φορολογικής αρχής και εταιρεία. Από την άλλη, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ευελιξίας για συγκεκριμένα πιο απτά στοιχεία και αυτό ε, δίνει σημαντικό πλεονέκτημα σε κάποιες επιχειρήσεις απέναντι σε άλλους τόπους ή άλλες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει προς το παρόν ουσιαστικά καμία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών. Επειδή δεν υπήρξε κανένα αίτημα από καμία πλευρά, <coughs> υπάρχει και το επιχείρημα πλήρους συμμόρφωσης με τους ε, γενικούς κανόνες, όμως αυτό είναι μια ευρύτατη ερμηνεία, υπερβολικά ευρεία. Είναι σχεδόν αδύνατον να εξετάσει κανείς το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών για λόγους που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο με βάση το οποίο θεσπίζονται και περιλαμβάνει πλήρη εμπιστευτικότητα. είναι αδύνατον να λάβει κανείς ε, συγκεκριμένα και γενικότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Και πολύ συχνά αναφέρεται το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κεντρική καταχώρηση και είναι μία απλή διοικητική πράξη. Επομένω, είτε καταχώρηση δεν υπάρχει, το μητρό αυτό ενδεχομένω δεν είναι διαθέσιμο, ή γίνεται με διαφορετικό τρόπο, διαφορετική διαδικασία και αυτή ήταν και μια γραπτή απάντηση που λάβαμε από το Λουξεμβούργο. Σε ευρύτερο πλαίσιο λοιπόν κατανοείται την κατάσταση που παρατηρούμε. Και εγώ προσωπικά έχω τη γνώμη ότι υπάρχει μία κινητικότητα, μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την οτροπία και τις, ε, των φορολογικών διοικήσεων, αλλά και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την πολιτική ευθύνη για αυτό το θέμα, με πολλά στοιχεία που συνεπιδρούν. Πρόσφατα είχαμε το LuxLeaks και όλες αυτές τις αποκαλύψεις και άλλες περιπτώσεις πιο παλιά με την επισήμαση των κακών κειμένων και η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως έχουμε και κινήσεις του G20 και διεργασίες στο πλαίσιο του ΩΣΑ. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ατμόσφαιρα αλλαγής, ένα τέτοιο κλίμα αλλαγής αλλά τώρα πόσο αυτό θα διαμορφωθεί στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο δεν είναι τόσο σαφές προς το παρόν. Αρκετές νομικές εντότητες αλλά και τα κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε έχουν αυτόνομους ε, φορείς που ε, εξετάζουν τα ζητήματα των ε, φορολογικών συμφωνιών, των rulings. Η Ιρλανδία ρητός ζήτησε να μην αναφερθούμε στις φορολογικές συμφωνίες γιατί έχουν ε, ένα γνωμοδοτικό όργανο, αλλά σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, κάτω χώρες, έχουμε αξιωματούχους, φορολογικούς αξιωματούχους υψηλού επίπεδου, που έχουν μερική ή και πλήρη ανεξαρτησία και δεσμεύονται και οι φορολογικές αρχές και όταν ρωτήσαμε τα κοινοβούλια στο βαθμό στον οποίο μπορούν να ελέγξουν τη δραστηριότητα αυτών των ε, υπηρεσιών, είδαμε ότι υπήρχε μια ευρύτατη ποικιλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ή τουλάχιστον οι αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, ελαμβάνουν ετήσια έκθεση ε, στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι αθροισμένα ή και ανώνυμα αλλά δεν εξετάζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιριών που καλύπτονται από ε, την επιστατικότητα. Οι πρακτικές που ακολουθούνται για την προσέλκυση επιχειρήσεων ποικίλουν Δεν χρειάζεται τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά αυτές τις επιμέρους πρακτικές, όμω Κάποια στοιχεία νομίζω ότι καλό είναι να τα αναφέρουμε σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση των μη συνεργάσιμων επικρατιών και δικαιοδοσιών. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα ασαφής ταξινόμηση. Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική γνώμη και παραπέμπει στον ΩΣΑ και τον αντίστοιχο κατάλογο των μη συνεργάσιμων ως ευρύτερο πλαίσιο. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις επιβεβαιώνεται ότι καμία δικαιοδοσία δεν είναι συνεργάσιμη ή ότι είναι λίγες οι οποίες γενικά συμμορφούνται, όμως υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Σε... Δεν ξέρουμε για... ακριβώς... γιατί ακριβώς μιλάμε και δεν έχουμε αντικειμενικά κριτήρια. Τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη επίσης ποικίλουν, όμως συνοπτικά μπορώ να πω ότι επικεντρώνεται περισσότερο στον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματο και όχι ε, στον ονομαστικό συντελεστή. Επομένω, ο υπολογισμό του ε, ονομαστικού συντελεστή είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολλαπλές ε, συμφωνίες διμερούς χαρακτήρα και βλέπουμε ότι κάποιες χώρες μπορούν να έχουν 70, 80, 100 τέτοιες διμερές ε, συμφωνίες. Που εν γέννη ακολουθούν το πνεύμα των κριτηρίων του ΩΣΑ, αυτό μας είπαν. Αλλά είναι ιδιαίτερα ασαφή όλα αυτά. Για τα παιδιά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, patent boxes, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, όμως και πάλι ασαφής είναι και αυτή η έννοια. για το κατά πόσον διάφορα στοιχεία γίνονται παραδεκτά, όπως το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο. Έχουμε τη γενική εντύπωση ότι η ανταλλαγή προφοριών για τις φορολογικές συμφωνίες είναι αποδεκτή και σημαντική, όμως και πάλι πρέπει να εξετάσουμε αν είναι θέμα δημόσιο ή όχι. Μετά, για τις εκθέσεις αναχώρα και πάλι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα, δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω. Για την κοινή ενωπημένη φορολογική βάση έχουμε μια γενική συνένεση, εφόσον βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απομακρυνθεί από την ε, τρέχουσα εκδοχή. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της ενοποίησης που θέτει και το ζήτημα της ε, τιμής μεταβίβασης. Με την εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου που είπε ρητός, αρνήθηκε αυτό το ενδεχόμενο και γενική συμφωνία και συνένεση ό,τι αφορά την εξέλιξη του ΒΕΠΣ του ΩΣΑ. Δεν θέλω να καταχαστώ περαιτέρω του χρόνου σας. Απλώς ήθελα να κάνω μια γενική αρχική σύνοψη των πορισμάτων μας. Αλλά θα μείνω εδώ. Δεν έχει έρθει ώρα να τα εξετάσουμε όλα αναλυτικά. Κάτι τελευταίο για την Ελβετία. Η διάδουσα περίπτωση. Στη σύνοψή μου εγώ αναφέρθηκα περισσότερο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερως ε, η περίπτωση της Ελβετίας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Εν μέρει οι συμφωνίες έγιναν βάσει μιας μελλοντική προσχώρησης, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολύ ιδιαίτερε λοιπόν σχέσεις ε, ειδικού περιεχομένου με την Ελβετία αλλά κάπου πάγωσαν τα πράγματα σε αυτή τη διαδικασία. Και τώρα είναι λίγο περίεργες οι σχέσεις μας, όμως δεν νομίζω ότι μπορούμε να το ε, εξετάσουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ Ελίζα. Μικάλ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε ορισμένε ακροάσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ακούσαμε μια σειρά από εμπειρογνώμονες και όπως μας είπε τώρα και η συνάδελφος ε, Ελίζα Φερέρα και ο Πρόεδρος, πήγαμε σε έξι χώρες. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να κάνουμε αυτές τις αναλυτικές ε, εργασίες. Διαπιστώνουμε, ωστόσο, ότι σε κάθε επίσκεψη, σε κάθε συζήτηση, μετά τις συζητήσεις προέκυψαν περαιτέρω ερωτήσεις που χρειάζονται περαιτέρω εξέταση. Να αρχίσω με το, με το θέμα συγγνώμη, αυτό που καταγγέλουν ε, παρανομίες, τον whistleblower. Ξέρω ότι όσοι το κάνουν αυτό, μετά υφίστανται τρομερές ε, συνέπειες. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει συνένεση μεταξύ μου ότι είναι επίγουσα ανάγκη να επανεξεταστεί η προστασία αυτών των καταγγελόντων. Είναι απόλυτα αναγκαίο. Δεν μπορούμε να δεχθούμε από ηθική πλευρά. Αυτοί που καταγγέλουν, για παράδειγμα, περιπτώσεις φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, κατόπιν, να αντιμετωπίζονται οι ίδιοι μέσω ποινικών διαδικασιών. Ενώ εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν τη φοροδιαφυγή, που στις περισσότερες χώρες είναι ποινικό αδίκημα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παθαίνουν τίποτα απολύτως. Δεν ε, ισχυρίζομαι βέβαια ότι η παροχή εμπιστευτικών εμπορικών στοιχείων στον τύπο θα πρέπει να είναι η καλύτερη μέθοδος, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ούτω ώστε στην Ένωση, σε όλα τα κράτη-μέλη, μέσω κάποιας δικαστικής συνεργασίας, για παράδειγμα, να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες καταγγελίες των whistleblower σε κρατικές αρχές που φτάνουν σε αυτές τις κρατικές αρχές και οδηγούν κατόπιν σε έρευνες να γίνονται σε καθεστώς προστασίας αυτών που κάνουν αυτές τις καταγγελίες. Να μην υφίστανται δηλαδή επιπτώσεις μετά. Να μην έχουν ε, τη μοίρα αυτών των οποίο εγώ διαπίστωσα και μου με συγκίνησε πολύ. Για παράδειγμα κάποιοι Γάλλοι που έκαναν καταγγελίες, ναι με δικαιώθηκαν στα δικαστήρια, αλλά έκτοτε δεν μπορούν να βρουν δουλειά πουθενά, διότι Κανένα επιχειρηματίας δεν θέλει να του προσλάβει. Επειδή έκανε αυτό που έκαναν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Αντιρρήσεις και συμφωνίες διαπιστώσαμε. Σε διάφορες χώρες οι συνάδελφοί μας των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και οι εμπειρογνώμονες πολύ ανοιχτά και σαφέστατα μας είπαν ναι, βλέπουμε ότι η κάθε χώρα προσπαθεί να κάνει πιο ελκυστική τη φορολογία της, αλλά μας είπαν ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι κάτι το δεκτό. Όλοι θέλουν να προσελκύσουν εταιρείε, κυρίω για τι μικρότερε χώρε ισχύει αυτό. Μα το είπαν οι μικρότερε χώρε ότι αν δεν υπάρχει κάποιο φορολογικό πλεονέκτημα, δεν θα πάει κανεί να κατασταθεί σε μια μικρή χώρα, άρα δεν θα έχει φορολογικά έσοδα. Άρα θα έχει πρόβλημα προπολογισμό τη χώρα. Σε σχέση με αυτό τίθεται βέβαια και το θέμα πώς ορίζουμε ένα μικρό κράτος μέλος. Για παράδειγμα στο Βέλγιο μας το είπαν αυτό και στην Ολλανδία, ότι είμαστε μικρές χώρες. Κατά τη χώρα μου δεν είναι και τόσο μικρές αυτές οι δύο χώρες. Θα έλεγα ότι είναι μεσαίων διαστάσεων. Άρα πρέπει να το δούμε και αυτό. Βεβαίως από πλευράς αρχής ε, δεν είναι ούτε παράνομο ούτε απορριπταίο ο φορολογικό ανταγωνισμό. Αλλά τι μπορεί να θεωρηθεί θεμητό φορολογικό ανταγωνισμό και τι επιθετικό ανταγωνισμό. Τι είναι αθέμητο. Και τι θα ήταν θεμητό και δίκαιο. Κατά τις επισκέψεις μας λοιπόν στην Ελβετία ακούσαμε τα εξής ενδιαφέροντα οι αντιδράσει, για να το πω διπλωματικά, δεν ήταν πάντα τόσο φιλικέ όταν εμεί βάλαμε το δάκτυλο στην πληγή. Όταν είπαμε, για παράδειγμα, όταν το καντόνι Βό, για παράδειγμα, που ισχύει και για άλλα καντόνια, όταν το καντόνι Βό, λοιπόν, δίνει εκπτώσεις φόρου σε κάποιες επιχειρήσεις, αλλά μόνο επιχειρήσει και μόνο για κέρδη, για κέρδη συγκεκριμένα, που έχουν προκύψει εκτός Ελβετίας. Τότε ακόμη και ο απλούστερος άνθρωπο καταλαβαίνει ότι στόχος αυτής της νομοθεσίας είναι να προσελκύσει ξένες εταιρείε. Βεβαίω η ελβετική κυβέρνηση έχει πει ότι μέχρι το 2017 θα έχει καταργηθεί αυτό, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει όχι μόνο στην Ελβετία αλλά και σε κράτη-μέλη της Ένωσης υπάρχουν τέτοιες πρακτικές. Δηλαδή διάφορες δομές που έχουν σαφή στόχο να προσελκύσουν επενδύσεις από το εξωτερικό. Αυτό που είναι θετικό στην Ελβετία είναι, ξέρετε ότι έχουν τα καντόνια φορολογική αυτονομία. Ήδη όμως από την δεκαετία του 50 καθορίστηκε ένα πλαίσιο για να υπάρχει στο εσωτερικό της Ελβετίας θεμητός ανταγωνισμός, δηλαδή μεταξύ των καντονίων. Και τέθησαν δύο ελάχιστες προϋποθέσεις. Πρώτον, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, δηλαδή επιμένει και επιβάλλει η Ελβετία μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών των καντονίων και της Ομοσπονδίας γίνεται ανταλλαγή στοιχείων. Οπότε η πρόταση της Κομισιόν για αυτόματη ανταλλαγή προφοριών δεν δημιουργεί πρόβλημα. Και αυτό που εισήγαγαν στο εσωτερικό τη Ελβετίας είναι η κοινή βάση του εταιρικού φόρου. Και αυτό ανταποκρίνεται στις προτάσεις της Κομισιόν. Όμως είναι λυπηρό ότι μάθαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν το υποστηρίζουν αυτό όλα. Η Ελίδα Φερέρα μίλησε για τον Υφυπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Secretary of the Treasury. Είπε ότι είναι ακόμη, έχουν αφιβολίες για την ε, κοινή ενοποιημένη βάση του εταιρικού φόρου, το CCCTB. Ο προηγούμενος πρόεδρος ε, της ε, Μόνιμης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου της Βουλής των Κοινοτήτων, η Μάργαρετ Χότζ, είχε πει ότι είχε ακούσει για ευνοικέ συμφωνίε μεταξύ της εφορίας, sweetheart deal τα λέγανε, και της επιχείρησης Goldman Sachs. Τώρα όμως μας ε, διαβεβαίωσαν οι φορολογικές αρχές ότι δεν υπάρχουν τέτοιες φορολογικές συμφωνίε, Το αναφέρω ως παράδειγμα. Ότι υπάρχουν ε, αντιφάσεις ε, σε αυτά που μας λένε, πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Άλλα δύο σημεία, συντόμως σε σχέση με αυτό πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και καινοτομίας για τα θέματα δηλαδή διανοητικών δικαιωμάτων. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποια είναι η οικονομική αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα για, ορισμένες, ε, για ορισμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να λάβουν διπλή αποζημίωση για τα έξοδα που έχουν κάνει για έρευνα και ανάπτυξη. Υπήρξαν πολύ έντονε συζητήσει για τα θέματα αυτά κατά την επίσκεψή μα ε, στην Ολλανδία. Και τελευταίο. Φορολογική παράδειση. Αν δούμε περιοχές όπως τα νησιά Guernsey, Jersey, Isle of Man, όλα αυτά στη μάχη, το Γιβραλτάρ, οι Παρθένες νήσου, οι, Βρετανικές Παρθένες νήσοι. Να δείτε τι ύψος επενδύσεων και κύκλου εργασιών διαπιστώνουμε σε αυτές τις χώρες. Είναι φανερό από την πρώτη ματιά ότι οι πόροι οι οποίοι εισέρχονται σε αυτές τις χώρες δεν είναι επενδύσεις στην ε, πραγματική οικονομία επενδύονται εκεί για να ξαναβγούν μετά σε άλλες πραγματικές οικονομίες. Οπότε θα πρέπει η Επιτροπή μας να το προσέξουμε αυτό. Να το προσέξει αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους προλογικούς παραδείσους. Η Ελίζα, ο πρόεδρος και εγώ, ε, άτυπα το συζητήσαμε. Μήπως δηλαδή θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε ως εξή σας ενημερώνω. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ενιαία αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Άρα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα. Υπάρχει αυτή η ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων, οπότε δεν μπορούν πάντα τα κράτη-μέλη να φορολογήσουν τα κεφάλαια από εκεί που προέρχονται. Μήπως λοιπόν στα εξωτερικά σύνορα τότε, τα φορολογικά εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, θα μπορούσαμε να υπάρχει κάποια μορφή ελέγχου ή φορολόγησης, ούτως ώστε να υπάρξει μια ισότητα. Γιατί όσοι υπάρχει διπλή μη φορολόγηση. Οι συμφωνίες διπλής φορολόγησης μπορεί να είναι μια λύση. Ακόμη και η πληρωμή μερισμάτων στις Ολλανδικές Αντίλες ή στο Τρινιτάρκετο και τον Τομπάγκο ή στα Μπαρμπέιντος έχουμε πολλά παραδείγματα και στο Λουξεμβούργο τα είδαμε πρέπει να εξεταστεί. Γιατί γίνονται σε αυτές οι μεταφορές μερισμάτων χωρίς να φορολογούνται. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μικαήλ. Ανλής Ντότς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα λίγα σχόλια. Συμφωνώ με τα περισσότερα που είπαν οι συνάδελφοι και νομίζω ότι οι συζητήσεις που είχαμε ε, στην Ειδική Επιτροπή θα βοηθήσουν πάρα πολύ και εμένα και τον κύριο Νίντε Μάιερ για να συντάξουμε την ε, έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας. Φυσικά έχουν γίνει πολλές εκκλήσεις από το Κοινοβούλιο στο παρελθόν για να βελτιώσουμε τους κανόνες για τον εταιρικό, την εταιρική φορολογία, αλλά μάθαμε και πολλές νέες πρακτικές και πολλά νέα προβλήματα που χρήζουν ε, νέων προβλημάτων για να αντιμετωπιστούν. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για τη δουλειά που έκανε οργανώντα αποστολέ αυτέ, επισκέψει αυτέ. Δύο σχόλια συγκεκριμένα. Καταρχά, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι δημόσιο, αλλά οι Βέλγοι προσπαθούν να αλλάξουν δεχομένω του κανόνε για τα υπερβολικά κέρδη. Θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα αυτή τη Επιτροπή, γιατί ζητήσαμε του Βέλγου και στην επίσκεψή μα πολλέ φορέ το θέμα αυτό να συζητηθεί και τους πιέσαμε γύρω από αυτό το θέμα. Ίσως λοιπόν, να, κάποια πρώτα αποτελέσματα από τις ερευνές μας. Για την περίπτωση του Βασιλείου. Δεν θα να είμαι άδικη, αλλά δεν κατάλαβα εάν ο Υπουργός ήξερε τις ε, λεπτομέρειες του πακέτου της Επιτροπής για το CDB όταν συζητήσαμε. Όταν συζητήσαμε με υπαλλήλους στην συνεχεία, το μήνυμα είναι ήταν διαφορετικό βεβαίως. Είπαν ότι τα στοιχεία της, του πακέτου της Επιτροπής για το CCTB που καλύπτουν τα μέτρα αντιμπέψ θα εξεταστούν με ανοιχτό πνεύμα. Και επαναλήφθηκε αυτό και στο υλικό που μας έδωσε η κυβέρνηση. Δεν θέλω να αφήσω αλόβητη και την ε, κυβέρνησή μου. Αναφέρθηκε αυτό το θέμα. Merci, Monsieur Viegas. Δεν ξέρω αν όλε οι εξαρτώμενε περιοχέ του θέματο ε, και αυτέ συμμορφώνονται με τα φορολογικά μέτρα. Ευχαριστώ. Για αυτές τις έρευνες θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή μας σεβάστηκε και έπαιξε μάλλον το ρόλο της που ήταν ποιος να συλλέξει πληροφορίες και να έρθει σε επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτό το πεδίο που είναι και περίπλοκο και πολυπίκυλο. Και αυτά που μαθαίνουμε, αυτά που μα δείχνουν τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Δεν μας εκκλείσει αυτό. Μετά από τι διάφορε επισκέψει, αυτό που προκύπτει από αυτέ τι επισκέψει ανεξάρτητα από την καλή θέληση που μπορεί να δείχνουν κάποιοι, κάποιοι φορείς και κάποιες αρχές, υπάρχει αυτή η ανησυχία για όλες τις χώρες που επισκεφτήκαμε. Δηλαδή, όλες αυτές οι χώρες πρέπει να ελέγξουν κάποιες επενδύσεις, να αποφύγουν ε, κάποιες επιχειρήσεις να μετεγκαθίστανται όσο μπορούν να τις αποτρέπουν. Φυσικά υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Ειδικά σε παγκόσμιο κλίμακα. Υπάρχει επίσης και ένας ολόκληρος κλάδος συμβούλων νομικών, φορολογικών συμβούλων, τεχνικοί ε, που δουλεύουν με τις επιχειρήσεις και δίνουν πληροφορίες πολύ πιο προηγμένες, ε, πολύ πιο ενδελεχείς από, ε, και είναι σε ένα επίπεδο πάντα πιο, πιο πάνω και πιο πέρα από αυτό που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις, οι δημόσιοι φορείς κτλ. Δεν ξέρω τώρα σε ποια επίσκεψη είχα σκεφτεί, το άκουσα αυτό, αλλά κάποιο είπε ότι τα πρότυπα του ΩΣΑ για τη διαφάνεια ε, για τον κύκλο εργασιών και τα λοιπά και για τα κέρδη είναι κενά περιεχομένου. Και ε, κάθε φορά οι σύμβουλοι είναι σε θέση να αποφεύγουν, να συμβουλεύουν τις εταιρείε για να αποφεύγουν ε, αυτά τα πρότυπα. Επίσης, η φορολογική παράδειση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Την αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει ένας κατάλογος χωρών που δεν συνεργάζεται. Ε, τελικά δεν έχει κανένα νόημα αυτός ο κατάλογος όμως, αφού τις αφήνουμε έτσι αυτές τις χώρες. Η δουλειά της Επιτροπής μας θα είναι να επιταχύνουμε και μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις της Επιτροπής βοηθούν γιατί είπαν, είπε η Επιτροπή ότι θέλει να δημιουργήσει ένα πιο επικυροποιημένο κατάλογο φορολογικών παραδείσων. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, πάνε προς σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα και τη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ στην ε, ειδική μας επιτροπή. Θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό κατάλογο χώρων που συνεργάζονται και που δεν συνεργάζονται. Θέλουμε να κάνουμε μια καταγραφή πιο ε, λεπτομερή. Θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε την παρουσία φορολογικών παραδείσων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει μεγαλύτερη συνείδηση αυτού του φαινομένου. Και κάτι άλλο το οποίο μου ε, μου έκανε εντύπωση και που είναι σημαντικό, είναι ε, μια ιδέα που προκύπτει από το Λουξεμβούργο. Δηλαδή η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές συμφωνίες, για τα tax ruling. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση. Γίνεται δεν γίνεται. Δηλαδή, μας είπαν, ναι, υπάρχει μια πληροφορία, εμείς διαβιβάσαμε αυτές τις πληροφορίες για αυτά τα, τις φορολογικές συμφωνίες, αλλά δεν δόθηκε καμία απάντηση. Α, εν αυτή περιπτώσει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να το, να το δώσουμε μεγάλη δημοσιότητα, να το δημοσιοποιήσουμε. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να δημοσιοποιείται εάν θέλουμε να ελοπίσουμε το στόχο που έχουμε θέσει. Και το τελευταίο θέμα. Αφαιρέθηκαν τρεις ή τέσσερις σελίδες για πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές και δεν φτάσαν στην Επιτροπή μας από μία έκθεση. Αυτή η έκθεση θα πρέπει, η έκθεση θα πρέπει να ε, δημοσιευθεί εν το συνόλο της. Δεν θα πρέπει να αφαιρούνται πληροφορίες που ενδεχομένως είναι πιο σημαντικές και που είναι αυτές που αφορούν τις δραστηριότητε ε, του Προέδρου Γιούνκερ. Μιλάω πάντα για την επίσκεψη στο Λουξεμβούργο. Ε, και ο Γιούνκερ θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στις εργασίες της Επιτροπής μας. Ας τον εμπλέξουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε για να χωρίς μικρόφωνο. Ήθελα να χαιρετήσω τις επισκέψεις αυτές και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που μας παρουσίασαν οι συνάδελφοι που συμμετείχαν σε αυτές τις επισκέψεις. Εγώ συγκρατώ το εξής. Πώς οι φορολογικές μας αρχές κάνουν αυτό το race to the bottom, όπως λέγεται. Ανταγωνίζονται δηλαδή η μία την άλλη για, τον, για τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Και αυτό μάλιστα παρουσιάζεται ως ε, κάτι πολύ φυσιολογικό. Ιδίως μετά την ε, θέσπιση του νέου νομίσματος. Γι' αυτό και τα συμπεράσματα που εμείς θα ε, βγάλουμε στην δική μας στο δικό μας έγγραφο είναι πολύ σημαντικά. Συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να επιστήσουμε και την προσοχή σε όσους ε, μας επέτρεψαν να τα ανακαλύψουμε όλα αυτά, τους λεγόμενους δηλαδή whistleblowers. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τη δική του σημασία και μάλιστα πολλοί έχουν διώκονται και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ήθελα λοιπόν να ζητήσω να μην ξεχνάμε τις περιπτώσεις κρατών μελών που δεν έχουν κατά πάσα πιθανότητα φορολογικές συμφωνίες, tax rulings, όμως έχουν άλλες αθέμητες πρακτικές και πολιτικές εγώ αναφέρομαι στη χώρα μου, αλλά σίγουρα δεν θα είναι και η μοναδική που υφίσταται ε, απίστευτα μέτρα λιτότητας και ανταπορριγωγικά από την Τρόικα κατά τη γνώμη μου, που δημιούργησε τεράστια φορολογική ανισότητα στους ε, φορολογουμένους, που πληρώνουν δηλαδή τους φόρους τους. Φόρους δηλαδή ατομικής ε, περιουσίας αύξηση φόρων για προσωπικών εισφορών που το 2012 ο Υπουργός Οικονομικών έλεγε ότι ήταν απαράδεκτη βάναυση αυτή η φόρη. Είχαμε ακόμα και πάνω από 50% δηλαδή φορολόγηση. Ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις έπαιρναν φοροαπαλλαγές, άλλα πλεονεκτήματα φορολογικά που για το 2013 ανέρχονται σε πάνω από ένα δις ευρώ με καμία απολύτως διαφάνεια και μάλιστα πορτογαλικές αρχές ή όταν ακόμα και υπήρχε υποχρέωση μάλλον για τις εταιρείες αυτές να δημοσιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία η υποχρέωση προς φορολογικές αρχές να δημοσιοποιήσουν τον κατάλογο αυτών των εταιριών δεν το έπραξε. Που είναι κάτι πραγματικά απαράδεκτο για... σε ό,τι αφορά την νομική και φορολογική δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, έχουμε και αυτή τη ζώνη της Μαδέρα, που είναι ουσιαστικά ε, φορολογικός παράδεισος. Και δεν ξέρουμε καν ποιε είναι οι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη ζώνη. Το ελάχιστο λοιπόν που πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο για μια χώρα που υπέστη ένα τέτοιο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από μερικά χρόνια ως επιτυχία, αλλά τελικά ε, μας οδήγησε σε αύξηση του δημοσίου χρέους, ε, επίπεδα μετανάστευσης που συγκρίνονται με την εποχή της δικτατορίας πριν από 50 χρόνια, με αυτή την μαζική μετανάστευση ατόμων με προσόντα, το brain drain όπως ονομάζεται. Και μια εξαιρετικά δυσάρεστη ε, προσαρμογή. Το ελάχιστο λοιπόν που μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο είναι αυτό. Και θα ήθελα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει εξηγήσει για τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών που έχει δημοσιοποιήσει. Και αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα αποτέλεσμα πολιτικών ε, διαπραγματεύσεων, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι δύσκολο να τα εξηγήσω όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Μπορούμε να θέσουμε αυτό το ερώτημα στον ίδιο τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα, Peter Simon. Για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της επίσκεψης στις διάφορες χώρες ήταν ότι συνήθως, δεν λέω πάντα, αλλά συνήθως όταν θέταμε το ερώτημα έχετε συνέστηση ότι κάτι δεν πάει καλά αντιμετωπίστηκα με άγνοια. Μου είπαν για παράδειγμα είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε πρώτες ύλες. Αυτό αξιοποιείται ως επιχείρημα ότι κάποιος χρειάζεται κάποιο ανταγων, ε, πλεονέκτημα ανταγωνισμού. Αλλά όταν εμείς κάναμε κάποια επικριτική παρατήρηση λέγοντας Μήπως αυτό είναι ε, αθέμητος ανταγωνισμός. Ποτέ δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Είπαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αθέμητος, αθέμητες μέθοδοι ανταγωνισμού. Ε, απάντησα πάντα η ανταγωνιστικότητα είναι αναγκαία. Οπότε εγώ εξάγω το εξή συμπέρασμα. Ότι ακόμη και αν καταφέρουμε να καταργήσουμε ορισμένες ε, μεθόδους, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν τη συμπεριφορά τους σε κάποιο άλλο επίπεδο με άλλες μεθόδους. Και αν το δει κανείς αυτό και το ε, αντιμετωπίσει και το αναγνωρίσει με απόλυτη ηρεμία, τότε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό που είναι απόλυτα αναγκαίο είναι η διαφάνεια. Χωρίς διαφάνεια δεν προχωράμε καθόλου. Πρέπει να ξέρουμε πώς γίνεται, ποιο holding αξιοποιείται, τι φορολογείται. Γιατί σε διάφορε χώρες είδαμε ότι 90% τη φορολογική βάσης υπολογίζεται με χαμηλό φορολογικό συντελεστή τότε τι έννοια έχουν οι χαμηλοί ή συγγνώμη οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστέ, εάν δεν υπάρχει διαφάνεια στο ποια είναι η φορολογική βάση. Αν τα έχουμε όλα αυτά, αν ξέρουμε ποιο πληρώνει πού και πόσα και ποιοι ειδικοί διακανονισμοί υπάρχουν και τι φορολογείται, ποια είναι η φορολογική βάση, τότε μόνο θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τη συζήτηση για τι σημαίνει δίκαιος ανταγωνισμός. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση όντως να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε και ποιος ακριβώς είναι ο στόχος μας. Στόχος μας είναι να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός και να υπάρχει για παράδειγμα μια δυνατότητα απόκλησης του ενός συντελεστή από τον άλλον. Αλλά πρέπει να γίνονται όλα αυτά με θεμητό και δίκαιο ανταγωνισμό. Αν δεν το επιτύχουμε αυτό, εάν λόγω της αντίδρασης κάποιων κρατών μελών για παράδειγμα. Εάν δεν υπάρξει ενοποιημένη βάση της φορολογικής βάσης, ενοποιημένη φορολογική βάση, εάν δεν έχουμε αναλυτική εικόνα για το ποιος που πόσα πληρώνει, τότε μπορώ να σας πω απόλυτα ήρεμα ότι η δική μου ε, απόλυτα υποκειμενική εκτίμηση είναι ότι δεν θεωρώ ότι μπορούμε να αλλάξουμε ουσιοδός τη συμπεριφορά των κρατών μελών. Διαφάνεια είναι η επίγουσα ανάγκη. Ευχαριστώ Πέτρα. Κάποια δικά μου σχόλια τώρα. Όπως είπαν και οι συγητές και πολλοί από εσά. κλείνει μια, τελειώνει μια εποχή. Σε κάποιες χώρες υπήρχε, όχι σε όλες, έτσι, υπήρχε μια περίοδος όπου κάθε κράτος θεωρούσε ότι μπορούσε να κάνει ό,τι του κάπνιζε για τα φορολογικά. Αυτή τη στιγμή οι υπόλοιποι δεν το παίρναν η ροδιά. Και κάποιες χώρες είχαν την τάση να θεωρούν ότι στην μεγάλη εσωτερική αγορά μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλαν, να είναι ελεύθεροι καβαλάριδες στα φορολογικά. Μερικές φορές οι ίδιε χώρες ή κάποιε άλλε χώρε καταχρώνταν της ευκολίας που υπήρχε να δανείζονται με χαμηλά ε, επιτόκια λόγω της ε, ένταξής του στο ευρώ. Υπήρχε αυτή ο ενθουσιασμός, αλλά κλείνει αυτή η σελίδα. Το LuxLeaks έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά το LuxLeaks δεν ήταν η πρώτη αποκάλυψη, μετά από, έγινε μετά από, από άλλες αποκαλύψεις, το offshore leaks κτλ τις Ηνωμένε Πολιτείε εδώ και δύο χρόνια συνέβη αυτό, σε άλλε χώρε ε, πέρυσι. Μέσω των συστάσεων του G20 και του ΩΣΑ, τα πνεύματα άρχισαν να αλλάζουν. Και βλέπουμε ότι σήμερα το πιο σημαντικό είναι το εξής. Και αυτό είναι, ισχύει για τις επιχειρήσεις, ισχύει για τα κράτη και για όλους όσους θέλουν να είναι χρηματοπιστωτικά κέντρα που ελκύουν διεθνώς τις εταιρείε. Η υπόλοιψη, η εμπιστοσύνη είναι βασικά πράγματα. Και η φήμη, καλή φήμη φτιάχνει κανείς να είναι σοβαρός. Ενώ παλιά όταν είχε την ικανότητα να ξεφεύγει. Αλλά τώρα η υπόλοιψη χτίζεται πάνω στη σοβαρότητα και για μας αυτό είναι το καλύτερο επιχείρημα ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι όπως υπόθηκε κιόλας ότι ενώ η λέξη ruling υπάρχει ε, στο κανονισμό της ειδικής μας επιτροπής στην πραγματικότητα ε, συμβολίζει την, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Ε, και μάλιστα λέμε ruling and other harmful practices, ε, συμφωνίες και άλλες επιζήμιες πρακτικές. Κάποιες συμφωνίες μόνο και πολλές άλλες πρακτικές όπως αυτή που είπε η Αναγκόμες στη χώρα της. αλλά εμείς βρήκαμε και άλλες πρακτικές και θα υπάρξουν και άλλες, πολλές άλλες. Και σε άλλες χώρες, πέρα από αυτές που επισκεφτήκαμε, που έχουν τέτοιες πρακτικές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, αυτό είναι προσωπικό μου, έτσι, ε, προσωπική παρατήρηση. Στις σχέσεις μας κυρίως με τα εθνικά κοινοβούλια που επισκεφτήκαμε. με, μέσω της εθνικής συνένεσης που δημιουργείται για να υπερασπιστούν οι χώρες τις εθνικές του ιδιαιτερότητες μεταξύ της ε, αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης συχνά. Ε, και ακόμα πιο εντυπωσιακό μεταξύ των ακαδημαϊκών, των εμπειρογνωμόνων που έχουν να αποδείξουν επιστημονικά και καλά ότι η χώρα τους έχει το πιο ουδέτερο, το πιο αντικειμενικό, το πιο ηθικό ε, σύστημα και το καλύτερο οικονομικά. Αυτό τα λέω έτσι για να σκεφτούμε λιγάκι βέβαια. Αλλά θα πρέπει αυτό να μας δείξει ότι παίζουμε καλά το ρόλο μας. Ότι με αυτόν τον τρόπο, τρόπο βοηθάμε όλους να αλλάξουμε κουλτούρα, να αλλάξουμε τα μυαλά του πονηρού, ε, του παμπόνηρου ε, και να περάσουμε από την κουλτούρα του, του ας πούμε, στην κουλτούρα του σοβαρού, του αξιόπιστου. Θα περιμένουν πολλά από εμά. Ο κόσμο ε, περιμένει πολλά από εμά, όχι μόνο για να κρίνουμε τα όσα συνέβησαν ε, τη δεκαετία 90, αλλά να δούμε ε, επί των βάσεων των όσων γίνονται τώρα, μετά το LuxLeaks, και στα κράτη που επισκεφτήκαμε, αλλά και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Οι φορολογικέ αρχέ και οι κυβερνήσει υποχρεώθηκαν να λάβουν υπόψη αυτέ τι αποκαλύψει και να αρχίσουν να αλλάζουν και την νομοθεσία τους και τις πρακτικές τους ή το ένα ή το άλλο τουλάχιστον ή και τα δύο ή το ένα ή το άλλο και στην Ελβετία ακόμα. Έτσι. Και εμείς, οι συγητές και εμείς μπορούμε να κρίνουμε αυτά τα πράγματα. Η Ελβετία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις φορολογικές συμφωνίες. Ε, διοικητικός πώς. Είναι η πρόοδος που θέλαμε. Η Ανλής μίλησε για το Βέλγιο. Οι Βέλγοι επίσης προσάρμοσαν την διοίκησή τους. Όταν πήγαμε να επισκεφτούμε το, τις βελγικές αρχές, ο φόρος για τα υπερβολικά κέρδη ίσχυε ακόμα. Και ήταν αντικείμενο επιχειρηματολογίες, επιχειρηματολογίας των φορολογικών αρχών. Ισχύει ακόμα αυτή η επιχειρηματολογία. Θεωρούμε ότι μια τέτοια νομοθεσία είναι αποδεκτή, γιατί είναι πολύ διάζουσα αυτή η φορολογία. Οι Ιρλανδοί θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταργήσουν το Double Irish, όλα τα προβλήματα εκλείπουν. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας ή άλλων χωρών, η κατάργηση και στην περίπτωση της Ολλανδίας, η μετατροπή των patent boxes σε innovation boxes Ε, το στάτους του, των ιδρυμάτων, των κληροδοτημάτων. των καταπιστευμάτων άλλαξε. Ε, μήπως κάναμε απλή αντικατάσταση ενός συστήματος με το, με όμοιό του. Εμείς πρέπει να το κρίνουμε αυτό, να κρίνουμε αν άλλαξε κάτι ουσιοδός. Και ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να τονίσω. την παραμονή της πολύ σημαντικής ακρόασης που θα έχουμε με την ΕΚΟΝ την επόμενη εβδομάδα και με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πιο επίπεδο, ε, το τελευταίο στοιχείο είναι ο επίγον χαρακτήρας. Τα Υπουργεία Οικονομικών έχουν απίστευτη ικανότητα να χρονοτριβούν. Επίσης, το κοινοτικό σύστημα έχει μια καταπληκτική ικανότητα να χάνει χρόνο. Να κερδίζει, να, πηγαίνει γρήγορα στην αρχή και να καθυστερεί μετά. Είμαι πεπισμένος ότι το κλειδί της επιτυχίας του Κοινοβουλίου μέσω των εργασιών της Επιτροπής Τάξ και των εργασιών της ΕΚΟΝ έγκυται στην ικανότητά μας να κρατήσουμε την πίεση, ούτω ώστε να γίνουν σημαντικότερες πολιτικές επιλογές φέτος επί Λουξεμβουργέζικης Προεδρίας. Και μάλιστα είμαι και αγωπημένος, ε, απογοητευμένος ε, προσωπικά από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι πολύ γενικόλογες και αόριστες και στο περιεχόμενό τους και ως προς το χρονοδιάγραμμά τους. Το χρονοδιάγραμμα είναι ένα στοιχείο κλειδί. Αυτό που δεν θα αποφασιστεί φέτος θα αποφασιστεί μετά από 20 χρόνια. Και το τονίζω αυτό γιατί εγώ τα ξέρω πολύ καλά αυτά, την ικανότητα που έχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα Υπουργεία Οικονομικών να αποφεύγουν τα προβλήματα, τα ακαθόδη, παραπέμποντάς τα στην επαύριο, περιμένοντας λέει ναι, μια ακόμα μελέτη, τις εκλογές που θα γίνουν στην ηχή χώρα, ε, διεθνείς ε, φορείς να μας κάνουν προτάσει προτάσεις κτλ. Η Ευρώπη προχωράει όταν βάζει καταληκτικέ ημερομηνίες, ατζέντα και αποφασίζει να σκοτωθεί για να σεβαστεί αυτές τις, ε, αυτές τις προθεσμίες. Ε, αυτό θα σκοτωθεί, έτσι, ε, είναι μια μεταφορά. Αλλά κοιτάξτε, επειδή μας έχει ασκεί υπογλυκαιμία και δεν έχουμε και άλλα θέματα στη μερίσια διάταξη, θα σταματήσουμε εδώ, θα ξαναπούμε στις 2 Ιουλίου για να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση με την ΕΚΟΝ και μέχρι τότε ενθαρρύνω τους εισηγητές μας που τους συγχαίρω κατά τα άλλα να συνεχίσουν τις εργασίες με τους σκιώδεις εισηγητές γιατί χρειαζόμαστε το σχέδιο έκθεσή τους το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ και λύεται εδώ η συνεδρίαση.